Σας παρακαλώ να αρχίσουμε να συνεδρίασει. 7 ε, συνάδελφοι είναι εδώ. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε μια συνεδρίαση των συντονιστών. Οι αποφάσεις είναι στα γραφεία σας με email που χθες το βράδυ. Αν δεν έχετε καμία παρατήρηση, κάντε την παρακαλώ. Εάν όχι, εντάξει. Περνάμε στη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Έχουμε τον κύριο Λόκεργκάτ, που είναι ο εισηγητής για το προπολογισμό και θα μας πει που, που έχουμε λήψεις. Μόρτεν, έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, Είχαμε αυτή τη συνάντηση χθε και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδης για τη συμμετοχή τους και νομίζω ότι δεν θα θεωρήσετε ότι θα υπερβάλλω αν σας πω ότι ήταν πολύ καλή η συνεδρίαση και νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι συνολικά υπήρξε ε, ευρεία συνένεση στην Επιτροπή όσον αφορά τα ζητήματα υποσυζήτηση. Βεβαίως είχαμε δύο θέματα εδώ. Είχαμε τη γνωμοδότηση για τις πολιτικές προτεραιότητες που ελπίζω ότι όλοι πήρατε και τις τροπολογίες στο σχέδιο προπολογισμού. Όπως ελέγχθη, επανειλημμένα, αλλά τώρα επιτρέψτε μου το επαναλάβω, στις 23 Ιουλίου έχουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες αυτές. Για να μην ε, το ξεχάσετε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ότι αν εξετάσουμε τη νέα διαδικασία, πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα αυτή τη φορά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Δεν έχουμε ένα δεύτερο γύρο και μόνο μία ρήψη, αν μπορώ να το πω. Αυτό βεβαίως περιπλέκει τα πράγματα, γιατί τώρα πρέπει να είμαστε λογικοί ευθύς εξ αρχής. Η νέα κατάσταση αποδεικνύει ότι το Συμβούλιο ε, έχει αναλάβει νέες αρμοδιότητες και θέλει να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές για να, για να προβεί σε περικοπές. Να μην σας επαναλάβω λοιπόν όλα τα αριθμητικά στοιχεία. Απλά και μόνο να πω δύο λόγια για ε, τους αριθμούς που αφορούν εμάς, αυτή την Επιτροπή. Οι περικοπές στο σχέδιο προπολογισμού θα είναι 25 εκατομμύρια στην ε, ε, μακροχρόνια ε, κατάρτιση 100 εκατομμύρια στους ανθρώπους, 8 εκατομμύρια του Erasmus Mundus και ε, ε, σχεδόν τα ίδια και στο ε, πολιτιστικό πρόγραμμα. Βλέπετε λοιπόν ότι τι γίνεται ακριβώς με τις περικοπές και τα, τα επιχειρήματα του Συμβουλίου φαίνεται ότι είναι ότι πρέπει να, κάνουμε το, πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, τακτική των κρατών μελών όσον αφορά τις περικοπές, περικοπές των ταπανών. Ναι, αλλά κατά την άποψή μου Αυτό δεν έχει καμία λογική. Υπάρχει μεγάλο χάσμα κατά την άποψή μου ανάμεσα στα ωραία λόγια που ακούμε και στις ε, στρατηγικές τις οποίες όλοι συμφωνούμε και μετά στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν βλέπω λογική στις περικοπές και μόλις χτες ε, είχαμε το Βέλγο Υπουργό, ο οποίο ήρθε εδώ και ο οποίο αναφέρθηκε σε αυτά, παρέμβασε σε μία πρόσφατη συνεδρία στη Μαδρίτη, όπου η Υπουργοί Παιδεία όλοι οι Υπουργοί Παιδείας συμφώνησαν ότι ε, χρειάζεται ένας ε, ε, σωστός προπολογισμό για να εφαρμοστεί η στρατηγική αυτή. Άρα δεν έχει λογική το όλο θέμα. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει μάστερ στα οικονομικά για να καταλάβει ότι αυτή η λογική ε, λείπει στη συγκεκριμένη περίπτωση και νομίζω θα πρέπει να εκφράσουμε τη διαφωνία μας έντονα συναντήθηκα με, το γενικό εισηγητή, με τη Γενική Εισηγήτρια, τη Συντόνια, και η άποψή τη είναι βεβαίω να αυξηθούν οι δεσμεύσει για την νεολαία, την εκπαίδευση και την κινητικότητα. Θεώρησε ότι οι περικοπές του Συμβουλίου αποτελούν πρόκληση, έτσι το έφεσε. Ε, λαμβάνοντα υπόψη προτεραιότητα στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα η συντόνια, η συντόνια χρειάζεται την υποστήριξή μα στη συγκεκριμένη περίπτωση και πιστεύω ότι πρέπει να τη δώσουμε την υποστήριξη αυτή. Όσον αφορά τη θέση μου, που φαίνεται το σχέδιο γνωμοδότησης, πρώτα απ' όλα, προτίθεμαι, όπως είπα και προηγουμένως, να αποκαταστήσουμε τον προπολογισμό όσον αφορά όλες τις περικοπές προτείνει το Συμβούλιο. Αυτό θέλω να προτείνω. Υποστηρίζουμε την Ευρώπη 2020 ε, μέσω του προπολογισμού 2011 και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι η εκπαίδευση είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία της στρατηγικής 2020. Άρα λοιπόν η διαβίου μάθηση, το Erasmus Mundus και, ε, το ε, People θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στη συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο προπολογισμό. Επίσης να αυξηθούν οι δεσμεύσεις για την επικοινωνία που αποτελεί σημείο κλειδί, όπως για παράδειγμα σε κρίσεις σαν αυτή. Όσοι ε, γνωρίζουν έστω και ελάχιστα στοιχεία για την επικοινωνία θα καταλάβουν αμέσω ότι δεν είναι η ώρα για να, περικο... για να προβούμε σε περικοπές στον προπολογισμό για την επικοινωνία. Αντίθετα, πρέπει να αυξήσουμε, ε, ε, αυξήσουμε την επικοινωνία σε τέτοιε στιγμέ. Δεν, λοιπόν, δεν έχουν λογική οι περικοπέ στο συγκεκριμένο θέμα. Επίση, θέλουμε να, να λοιπόν, να αυξηθούν οι οι πιστώσεις για την ε, ε, επικοινωνία. Να αυξούν τα κονδύλια για το θέμα αυτό. Και επίση όσον αφορά το θέμα τη κινητικότητα στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υποστηρίξουμε ε, τη δημιουργία αυτών των τριών νέων ευρωπαϊκών δημοσίων χώρων. Να αυξηθεί επίσης αυξήσεις και εδώ νομίζω ότι η χτεσινή συζήτηση αντικατοπτρίζει αυτή την επιθυμία και νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία και συνένεση στο συγκεκριμένο ζήτημα να αυξηθούν λοιπόν τα κονδύλια για τον αθλητισμό. Τα περιθώρια όμως είναι πολύ στενά αυτή τη φορά. Για να επαναλάβω τα νούμερα, στον τίτλο 1α 15,1 εκατομμύρια είναι το περιθώριο και στο 3β μόλις 15,2 εκατομμύρια. Άρα δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο λιγμών. Κάτι άλλο το οποίο θα προτείνουμε είναι ότι ακριβώς επειδή έχουμε το, το στενά περιθώριο για το 3β, το, το θα θέλουμε να το βάλουμε πάλι στο 4 για να δώσουμε περισσότερη άνεση στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη γραμμή. Όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προσκευαστικές ε, δράσεις, Πήραμε τα σχόλια από την Επιτροπή και οι προτάσει των μελών τώρα αποτελούν το κείμενο αξιολόγηση από την Επιτροπή και βαθμολογούνται με τους βαθμούς A, B, C, D, E. Θα τα είδατε αυτά. Και στη συνεδρίαση με τον Γενικό Διευθυντή είδαμε ότι υπάρχει επιθυμία για να εστιάσουμε την προσοχή μας στην σκοπιμότητα ε, κατά την αξιολόγηση ενώ των σχεδίων αυτών. Άρα δεν θα πρέπει να ε, ζητάμε να δοθούν κονδύλια για, μη, για ανέφικτα προγράμματα και σχέδια. Να συνεχίσουμε λοιπόν την εργασία μα ε, για τα προγράμματα που πήραν βαθμό A, B και C, Α, Β και Γ. Αυτή είναι η πρότασή μου και θέλω τι παρατηρήσει σα. Τελειώνοντας με το πρώτο τμήμα, να θέσω ένα ερώτημα προς το Συμβούλιο, που βρίσκονται εδώ. Φαντάζομαι τουλάχιστον δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Από ό,τι κατάλαβα, προτίθεστε να προτείνετε ε, προπαρασκευαστικές δράσεις ε, για ένα σημαντικό ζήτημα όσον, αφορά τους, ε, ε, τα, μνημεία. και βέβαια εδώ πρέπει να δούμε και το θέμα της νομικής βάσης. Της νομικής βάσης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί βρίσκεται στι προπαρασκευαστικέ δράσει το ζήτημα αυτό αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου όσον αφορά τα ποσά. 4 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται. Ε, μεγάλο αυτό το ποσό στο 3β που όπω σας είπα έχει περιθώριο μόλις 15,2 εκατομμύρια. Αυτά ήθελα να πω τώρα και βεβαίω ε, περιμένω τι ερωτήσει σας και τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Thank you, Martin. Ευχαριστώ πολύ Μόρτεν. Νομίζω είναι λυπηρό. Καταλαβαίνω, μίλησα με τον συνάδελφο Σάιτερ. Μου φαίνεται κατανόητο. στι δημοσιονομικές προβλέψει, πριν από τέσσερα χρόνια, αγωνιστήκαμε για να έχουμε περισσότερα χρήματα για την παιδεία και την πολιτισμό συμφωνήσαμε στις δημοσιονομικές προβλέψεις όταν μας έδισε περισσότερα χρήματα για αυτούς τους τομείς, παιδεία και απελεσμό το Συμβούλιο. Τώρα, η κατάσταση είναι η εξής. Ακριβώς σε το τον τομέα γίνονται περικοπές. Και δεν είναι επειδή δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα όπως στη Γεωργία, στο περιφορικό ή στο διορθωτικό ταμείο. 100% απορροφούνται τα κονδύλια αυτά και ζητούν για ακόμα περισσότερα μάλιστα. Και δεν καταλαβαίνω. Εκείνοι που τα εξετάσανε στο Συμβούλιο, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα. Και αν ένας ξεκινήσει με ένα σχέδιο, ίσως χρειάζεται λίγα χρήματα το πρώτο έτος, περισσότερα το δεύτερο και τα υπόλοιπα το τρίτο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αξιόπιστοι. Δεν μπορώ να εγκρίνω ένα σχέδιο για χι χρόνια και στο τέλος να μην δώσω αυτά που είχαν προβλεφθεί, που είχαν δεσμευθεί αν θέλετε. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από τα δημοσιονομικά, αλλά πραγματικά με σοκάρει αυτή η συμπεριφορά. Ταυτόχρονα όλοι λένε πολύ σημαντική η παιδεία, όλοι ξέρουν ότι στις περιόδους κρίσης και ο πολιτισμός είναι όσο πάει και πιο ε, σημαντικός και εδώ μας περικόπτουνε. Ανοησίες. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε από κοινού, μαζί με το Συμβούλιο, που ήταν πολύ αισιόδοξο χθε ο εκπρόσωπο, αλλά είναι ένα από του 27. Αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη, οι άλλοι κρύβονται πίσω από του Υπουργού Οικονομικών. Και μετά έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε νέε τροπολογίε. Και δεν μπορώ να πω θα πάμε στην κατηγορία της Κομισιόν ή όχι, γιατί μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες. Δεν είμαι και σίγουρη ότι οι ιδέες της Κομισιόν είναι σύμφωνες με τις δικές μας, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να επιλέξουμε εδώ πράγματα τα οποία είναι ορατά και έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τους πολίτες. Προσεγγίζουν τους πολίτες, γι' αυτό θα πρέπει να οχηθούμε. Ωραία. Ο Μάρκο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τη Μαρτίνα για το πλαίσιο που μας έδωσε. Θα ήθελα να επιστήσω λίγο την προσοχή σας σε ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό. Καταρχάς υπάρχουν ε, δύο απόψεις εδώ. Από τη μία πλευρά σε περίοδο κρίσης οι πολιτισμικές υπηρεσίες είναι οι μόνες οι οποίες εξακολουθούν να εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη. Άρα πρέπει να διατηρηθεί η πολιτισμική πολιτική των κρατών μελών γιατί είναι μία απάντηση προς την κρίση. Άρα οι περικοπές είναι παράλογες ειδικά σε προγράμματα που λειτουργούν καλά όπως στην εκπαίδευση. Επίσης, ε, ενώ υποτίθεται ότι για τον προϋπολογισμό αυτό δίνεται προτεραιότητα στους νέους, έχουμε περικοπές σε προγράμματα που αφορούν τους νέους. Για όλα αυτά πρέπει να πολεμήσουμε και χαίρομαι γιατί βλέπω την συγγήτρια να είναι αρκετά αποφασισμένη και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πολεμήσουμε αυτές τις περικοπές που κατά τη γνώμη μας είναι πρόκληση. Πρέπει λοιπόν να επανέλθουν οι προβλεπόμενες πιστώσεις. Και για να δούμε και θα έπρεπε να δούμε και ακριβώς τι σημαίνουν στην πράξη για τους νέους αυτές οι περικοπές. Τώρα, για τον αθλητισμό. Συνάδελφοι όπως ε, κύριε Μπελέ και Σαντιάγο έχουν αναφερθεί στο θέμα και εκεί πρέπει να αντιταχθούμε στις περικοπές. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μία συνάντηση με εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όσους λαμβάνουν δηλαδή τις αποφάσεις, γιατί πραγματικά δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με τις περικοπές που βλέπω στον πολιτισμό, στην διαβίω εκπαίδευση και στον αθλητισμό σε μία περίοδο κρίσης και ενδεχομένως θα έπρεπε να ζητήσουμε όχι διατήρηση των κοντιλίων, αλλά αύξησή του. Ευχαριστώ, Μόρτεν, για τις προσπάθειές σου Συμφωνώ και με τον προηγούμενο μιλητή. Όντως πρόκειται για πρόκληση σε περίοδο κρίσης ε, η μείωση αυτή του προϋπολογισμού. Προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε μεγάλα χρηματικά ποσά αγνοώντας τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, αν πρόκειται για πρόκληση, τότε και εμεί θα πρέπει να προκαλέσουμε και να ψηφίσουμε κατά τον προπολογισμό ομόφωνα. σω αυτή είναι μια λύση. Ε, για, να καταλάβουν τι κάνουμε. Διαφορετικά κανεί δεν καταλάβει τι κάνουμε. Ε, τι είμαστε, δηλαδή, μια επιτροπή για να μιλάμε ε, και το μόνο που κάνουμε είναι σε τελευταία ανάλυση ε, να σχολιάζουμε μια σειρά από θέματα χωρί να μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση. Νομίζω πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί. Vielen Dank. Bitte kurz fassen. Σα παρακαλώ, παρακαλώ, έστε σύντομοι. Δεν θέλουμε να συνεδριάσουμε το απόγευμα, θέλουμε να λύσουμε το πρωί. Παρακαλώ. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομη γιατί δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πρόκληση είναι η σωστή, η σωστή γιατί έπασε νομίζω. Και θα ήταν καλό ίσω στην γνωμοδότηση, όχι στο κονδύλι του προβολισμού, να πούμε ξεκάθαρα ότι βρίσκουμε απόλυτα απαράδεκτες περικοπές στον τομέα παιδείας και πολιτισμού και δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε πανηγυρικούς λόγους να εκθέτουμε την ε, να εκθεάζουμε την ε, σημασία των ποδία και του πολιτισμού και μετά να περικόπουμε τα κονδύλια. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό τη συγγνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Σύντομα, παρακαλώ. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος να πω ότι χτες με τον Μόρταν είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση. Συζητήσαμε τα θέματα του προϋπολογισμού και συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες ειδικά στο θέμα της διαβίου μάθησης είναι πρόκληση οι περίκοπες και πρόκειται να καταθέσουμε και τροπολογία για αυτό το θέμα καθώς και για τον αθλητισμό όπως είπε ο κύριος Φίσας επίσης ίσως θα έπρεπε να μην καταθέσουμε τροπολογίες αλλά να καταψηφίσουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα Όσον αφορά τώρα τους νέους, δεν είμαστε υπέρ μιας ειδική γραμμής του προϋπολογισμού και δεν ξέρουμε αν αυτό πρέπει να μπει σε, στη γνωμοδότηση σε τροπολογία. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μια, ένα κονδύλιο κατά, ή μια γραμμή τέλο πάντων κατά της ωραία, ναι, εν κινήσει. Δηλαδή, αν κάποιος πει κάτι έτσι άσχημο, αν υπάρχει κάτι σχετικό στην έκθεσή σου, μόνο το παρακαλώ να το διαγράψεις γιατί θα το καταψηφίσουμε αλλιώς. Η κυρία Κλάκη. Um, να κάνω δύο ε, σχόλια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικέ οι περιστάσει και ε, ευθύνη μα είναι να φροντίσουμε έτσι ώστε να πανώνται σωστά τα χρήματα φορολογουμένων. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Δεν είναι ότι εγώ δεν δίνω αξία στον πολιτισμό και στην ε, παιδεία, αλλά πρέπει να δούμε πού πραγματικά επιφέρουμε προσθέμενη αξία και να συντονίσουμε τα αποτελέσματα. Και κάτι το οποίο ήθελα να πω αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία, όπου ε, ο Γενικό ε, Γραμματέα εδώ ε, ε, βλέπει ότι κοστίζει 8,7 εκατομμύρια η όλη υπόθεση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ακριβώ. Πρέπει να επενδύσουμε και να αυξήσουμε τα κονδύλια στην έρευνα και στην εκπαίδευση, αλλά πρέπει να δείξουμε και μια κάποια μετριοπάθεια και να μην είμαστε άπλιστοι, γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Ähm, ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα βουλγαρικά. Θα ήθελα να σας πω ότι ο συνάδελφός μου που αναπληρώνω δεν μπορούσε να είναι παρόν. Θα σας πω δύο λόγια όσον αφορά το πρόγραμμα του για το ε, εκπαίδευση στα δεύτερα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από ό,τι άκουσα αυτό, είναι κάτι που είναι θέμα των κρατών μελών και δεν μπορεί να ενισχυθεί από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Εμείς δεν συμφωνούμε όμως με την Κομισιόν πάνω στην άποψή της αυτή, γιατί μπορεί αυτό να δώσει ίσως κάποια κίνητρα στα κράτη-μέλη και έτσι μπορούν έτσι και τα κράτη-μέλη να κινητοποιηθούν για να εισαγάγουν κάποια εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό τομέα μέσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καμιά φορά κάτι γίνεται. Εγώ δεν θα σας πω γιατί είναι σημαντική η παιδεία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Έχουμε κάθε συμφέρον οι νέοι να γνωρίζουν περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την ιστορία του, του θεσμικού του όργανα, την ε, νομοθετησία της. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, μπορούμε να αναλάβουμε κάποια βήματα ούτω ώστε αυτό το πρόγραμμα να προσαρτηθεί σε κάποια από τα ισχύοντα πρόγραμμα παρόλη την άποψη της Κομισιόν. Ίσως η δική μας Επιτροπή να μπορεί να προετοιμάσει μια έκθεση πρωτοβουλία σας παρακαλώ Πρόεδρε, λάβετε το και αυτό υπόψη Ωραία. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Μόρτεν που τόνισε τα βασικά σημεία της πολιτικής μας. Σε αυτή την περίοδο κρίσης οι περικοπές γίνονται παντού αλλά πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του πολιτισμού όπως είπε και η Μονίκ. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά αυτά που κάνουμε εδώ, το είπε και ο Σαντιάγο. Πρέπει πάντως να δούμε τι περιθώριο ελιγμών έχουμε πρώτη φορά ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ψαλίδα εντός της οποία πρέπει να κινηθούμε. Αν έχουμε κάποια περιθώρια ή όχι. Πάντως πρέπει να αντισταθούμε γιατί αυτοί που θα αντισταθούν περισσότερο ίσως θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν τα περισσότερα περιθώρια ελιγμών. Κοιτάξτε, Μαρή Εγώ συγχύζομαι πάντα αν κάποιος λέει τι είπε ο Ζώμονε. Εγώ ήμουνα δασκάλα και να σας τα πω τα πράγματα ξεκάθαρα. Ο Ζαμονέ δεν μπορεί να είπε τίποτε τέτοιο. Ήθελε να ενώσει άνθρακα και χάλιβα, οικονομία, τίποτα άλλο. Η ιδέα που οδήγησε περισσότερα ήταν ο Ρόμπερ Σούμαν. Και ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είπε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός υπάρχει, δεν χρειάζεται να, ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό που ε, οδήγησε στον πόλεμο για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Λοιπόν, το είπα πολλέ φορέ. Σα παρακαλώ όμω και εδώ το λέω να μην λέμε στη δική μα επιτροπή εδώ αυτά τα πράγματα που δεν είναι σωστά. Η κυρία Φεράν, κοιτάξτε, τα περισσότερα έχουν ελεγχθεί, θα είμαι σύντομη. Ε, είναι σημαντικό εδώ στην Επιτροπή να εκφράσουμε να πιστεύω για την παιδεία και τον πολιτισμό και σημαντικό είναι όμως ότι και οι συνάδελφοι από τις συναμόδιες επιτροπές ε, να θυμηθούν τι λέμε πάντα. Δεν μπορούμε από τη μια μεριά να μιλάμε για την ε, Ατζέντα 2020 όπου το 40% θα πρέπει να είναι από αυτή τη δευτοβάθμια σε εκπαίδευση, αν όχι τριτοβάθμια, και από την άλλη μεριά να μιλάμε εδώ για περικοπέ. Δηλαδή, άλλα λέω σήμερα, άλλα λέω αύριο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Και κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι σίγουρα έχει νόημα η επικοινωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο ειδικά και η Κομισιόν πρέπει να ξανασκεφτεί ούτως ώστε αυτό που ε, τυπώνουμε ή που εκδίδουμε να είναι λογικό. Αλλά ακριβώς την εκπαίδευση των δημοσιογράφων είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλοί ε, δημοσιογράφοι ιδίως στις τοπικές εφημερίδες δεν έχουν ιδέα το τι γίνεται εδώ και δεν παρουσιάζουν και τίποτα. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που θα πρέπει να αποστείλουμε. Υπάρχει συνέχεια να το τονίσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ κυρία Μπατία. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να επαναλάβω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, συμφωνώ απόλυτα και αυτό που θα ήθελα είναι να κάνω κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Γιατί πιστεύω ότι, ε, κοιτάξτε, εμεί δεν, πρέπει να αντιδράμε, πρέπει να ε, απαντήσουμε συγκεκριμένη δράση. Ε, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είμαστε μάρτυρε, έτσι. Ε, ήταν η επιτάση. Πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να λύσουμε τα πράγματα ε, και να τα ρυθμίσουμε. Δύο-τρία πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μια επιστολή, κάτι, ένα έγγραφο με τη θέση μα, υποστηρίζοντα αυτά τα οποία είπαμε και εδώ. Και ε, κάθε ένας από εμά να έρθει σε επαφή με ε, τον Υπουργό, ε, τον αρμόδιο στη χώρα του, να του πει τι ακριβώς γίνεται και κατά πόσα μας υποστηρίζουν ή όχι. Γιατί σε τελευταία ανάλυση τι είναι το Συμβούλιο. Είναι όλοι οι Υπουργοί Παιδείας, έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Άρα να μιλήσουμε με τους Υπουργούς Παιδείας της χώρας μας. Γιατί ε, όταν έρχονται εδώ φαίνεται ότι συμφωνούν μαζί μας Και μάλιστα μας έχουν δώσει πολύ υποστήριξη και περιθώριο στην Επιτροπή μας. Επίσης, να μιλήσουμε και να αποστείλουμε αυτή την επιστολή ε, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, πολιτιστικού φορεί, ε, συλλόγου γονέων, συλλόγους νέων, να πούμε, κοιτάξτε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Εμεί πιστεύουμε Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει, ότι υπάρχει κρίση και δεν πρόκειται να ζητήσουμε αύξηση του προπολογισμού. Τώρα, οι περικοπέ δεν έχουν νόημα. Γιατί ε, αν θέλουμε να μιλάμε για τους συγκεκριμένους στόχους, εκπαίδευση, καινοτομία, κατάρτιση και καταλαβαίνετε θέλω να πω, να κάνουμε έτσι μια κάποια φασαρία, ε, ε, να, να τραβήξουμε τη, ε, την προσοχή της κοινή γνώμης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα πρότεινα λοιπόν να κάνουμε μια κάποια τέτοια δράση. Παντά, αντί να πούμε θα καταψηφίσουμε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όχι από τώρα τουλάχιστον να, ε, ε, ε, να, να, να ταράξουμε κάπως τα νερά. Αυτό, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, κλείθηκε η επανάσταση, έτσι. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι διακοπές στις πατρίδες μας, στα σχολεία δεν είναι κανένας. Θα πρέπει το Σεπτέμβριο να έχουμε όμως την πρόταση. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε μπορούμε να τους συγχύσουμε όλους προσπαθώντας στις ε, εθνικές οργανώσεις να ανακοινήσουμε τα πράγματα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό μετά ίσως. Τι ας έχουμε. Μπίσκι. Ε, ότι πρόκειται να γίνουν περικοπές ε, στην πολιτισμό Λιπηλό, ότι πρόκειται να γίνουν περικοπές στην παιδεία, είναι δημόσια απάτη απάτη της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης, γιατί στη στρατηγική του 2020 αναφέρεται η παιδεία. Και το τονίζω αυτό. Εδώ έχουμε μία δημόσια απάτη. Πρέπει να το πούμε να το ξαναπούμε. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε περικοπέ στην παιδεία. Δεν θέλω η Ευρώπη να έχει ένα μουσείο στο μέλλον. Να δαπανεί λίγο πολύ ό,τι δαπανεί η Μαλαισία και η Κίνα ε, σε ποσοστό του ΕΠ. Πρόεδρος, ναι. Το πρόγραμμα είναι όμως ότι τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην ε, παιδεία φαίνονται μετά τις επόμενες, μετά τις πεθεμόμενες εκλογές και οι περισσότεροι συνάδελφοι σκέφτονται μόνο μέχρι τις επόμενες ε, εκλογές. Ανθρώπινο είναι, δυστυχώς, αλλά πρέπει να το πούμε και δημόσια πάτη, ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία έκφραση. Συνάδελφος Ράναρ. Πάρα πολύ σύντομα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το επιχείρημα ότι δεν επιτρέπεται ενώ έχουμε νέες αρμοδιότητες μέσω ε, του συνθήκη του Λισαβόνας το ανακοινώνουμε με χαρά στα κράτη-μέλη και δεν έχουμε μετά χρήματα ούτε να κάνουμε το πιο βασικό. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει ο καθένας και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Γιατί πραγματικά είναι παράλογο να έχουμε αρμοδιότητες και να μην έχουμε χρήματα για να πούμε ούτε ένα κέχι. Πρόεδρος, ναι, ευχαριστώ ενώ μάλιστα που μέχρι στιγμής χωρίς νομική βάση δαπανούσαμε χρήματα για τον λογισμό περισσότερα από ό,τι πρέπει να δαπανίσουμε τώρα. Τελείω απαράδεκτο και ακατανόητο. Ο κύριο Σβέρ. Κυρία Πρόεδρε, για τον προϋπολογισμό θα ήθελα να πω ότι αυτό το μήνυμα είναι αρνητικό και για τα κράτη-μέλη, γιατί εξαιτίας της κρίσης και τα κράτη-μέλη θα μειώσουν τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Και στέλνουμε ένα μήνυμα για την τάση που θα επικρατήσει και στα κράτη-μέλη κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Τώρα έχουμε την Κομισιόν. Κύριε Νάουτς, παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, Πρώτα απ' όλα θα είμαι σύντομο, αλλά θέλω να σα ευχαριστήσω για την υποστήριξη προς τις προτάσεις μας και να σας πω ότι ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις προτινόμενες περικοπές ε, από το Συμβούλιο για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνούμε από πολιτική άποψη αυτά τα προγράμματα σαφώ υποστηρίζουν την Ευρώπη 2020 και άρα θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε και όχι να τα περικόψουμε, αλλά και από τεχνική άποψη θα έχουμε πολλά προβλήματα με αυτά τα οποία προτείνει το Συμβούλιο. Ορισμένε από τις περικοπές που πληρώνει ε, στις διοικητικές ε, γραμμές, στην ουσία, ε, στην πράξη σημαίνουν ότι δεν θα μπορέσουμε πλέον να εφαρμόσουμε ορισμένα προγράμματα. Ένα παράδειγμα το EIT, ε, που είναι μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία. Προτείνουν να διατηρήσουμε τον προπολογισμό στο επίπεδο του 2010. Το EIT είναι ένα αυξανόμενο οργανισμό που θα πρέπει να ε, οικοδομήσει ε, συγκεκριμένε υπηρεσίε. Εάν γίνει αυτό που προτείνει το Συμβούλιο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεύτερον, αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε και από εσά, κυρία Πρόεδρε, οι περικοπές όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Σε όλες τις γραμμές βασικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να ε, εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε αναλάβει δεσμεύσει, έχουμε πολιτεί προσχέδια και προγράμματα όπω και εσεί είπατε. Άρα, μέχρι το τέλο του χρόνου δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα να πληρώσουμε αυτά τα οποία θα οφείλουμε. Άρα, θα καθυστερήσουμε τι πληρωμέ, ε, θα πληρώσουμε επιτόκια στι ε, καθυστερήσει κτλ. Δεν θα εξοικονομήσουμε λοιπόν χρήματα, θα μα κοστίσουν περισσότερο όλα αυτά. Άρα, δεν έχει νόημα αυτή όλη η ιστορία. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ σύντομα. Ε, συμφωνούμε με ε, την ε, άποψη του εισηγητή όσον αφορά την επικοινωνία. Νομίζω ότι ήμασταν πιο τυχεροί από μεριά επικοινωνία έναντι της εκπαίδευσης. Μόλις 1,5 εκατομμύριο μας μείωσαν όσον αφορά τις, μείωσαν τις πιστώσεις πληρωμών, αλλά ισχύουν τέτοια επιχειρήματα που ισχύουν εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τώρα δεν ξέρω θα πρέπει να το αναφέρω τώρα αυτό το θέμα. Άρα, αλλά ε, πρότεινε το Συμβούλιο στον προπολογισμό μας να αυξηθεί ο προπολογισμό μα κατά 4 εκατομμύρια, παράδοξο αυτό, για να υποστηριχθεί το Ίδρυμα Auschwitz ε, ε, ως, ε, ως ένα είδος προπαρασκευαστικής δράσης που θα συμπεριληφθεί στα πλαίσια του συνολικού προγράμματος της Ευρώπης για τους πολίτες. Ε, το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά αν υποστηρίξετε μια τέτοια αύξηση, τότε νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Έχουμε και άλλα δύο συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την επικοινωνία, πέραν αυτών που αναφέρθηκαν ήδη, του ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, όπου με τη δική σα συμφωνία θέλουμε να ανοίξουμε άλλου τρει θα κοστίσει λίγο παραπάνω χρήματα αυτό το θέμα. Και τρίτον, θέλουμε περισσότερα, λίγο περισσότερα χρήματα στα δίκτυά μας για να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες συντονισμού και στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτά τα ανέφερε όμως και ο Μόρτεν και με την υποστήριξή σας θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για ε, να ε, μεταφέρουμε καλύτερα το μήνυμα της Ευρώπης και των δραστηριοτήτων στους πολίτες και να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της Ευρώπης και των πολιτών. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, we are. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναδώσω το λόγο στον Μάρτιν. Αλλά όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τουλάχιστον την πρόταση της Κομισιόν. Για τον προπολογισμό εννοώ. Ξέρει τι πρέπει να δαπανίσει, τι έχει υποσχεθεί, που έχει δεσμευθεί και εκεί που δεν μπορεί να πληρώσει θα αναγκαστεί να πληρώσει και τόκους γιατί θα πληρώσει αργότερα είμαι έξαλλη κυριολεκτικά πιστεύω ότι το Συμβούλιο πάει πραγματικά να μας εξαπατήσει τελείως και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα εκτός μικροφώνου δυστυχώς το Συμβούλιο ήταν, είχε έρθει χθες. Είχε έρθει χθε. Εσύ δεν ήρθε. Ήρθε το Συμβούλιο και μας υποσχέθηκε λαγούς με πετραχίλια χτες. Τι να κάνει όμως. Ε, νομίζω ότι οι πραγματικά έτσι σκέπτονται όπως μας είπανε. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άλλοι 26. Από τους οποίους υπάρχουν και μεγάλοι έτσι ογκώδεις και είπανε δεν τρέχει τίποτα, εμείς θα περικόψουμε. Ίσως είναι μια απειλή ίσως ξέρουν ότι εμείς δεν θα δεχθούμε τις περικοπές και θα μπορέσουν έτσι να τα πάρουν από αλλού. Τι να σας πω. Δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι τους, οπωσδήποτε. Θα πρέπει να εκφραστούμε έντονα και αν διαδιαφωνείτε εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής θα αποστείλω επιστολές σε όλες τις κυβερνήσεις της Ένωσης και θα τους πω ότι εδώ πραγματικά αυτοεξαπατούνται. Και τι είπαμε, δημόσια απάτη, δημόσια απάτη, ναι, πολύ ωραία. Δεν θα πω ότι είναι του κυρίου Μπίση γιατί άλλως θα με κυνηγήσουν στη χώρα μου. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι καλή η διατύπωση και θα τη χρησιμοποιήσω. Ναι, εντάξει, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ στη Γερμανία πρέπει να είμαι προσεκτική, ε. Δεν πρέπει να αναφέρουμε πάντα τον Εφευρέτη και η συνάδελφος ανέφερε τον λάθος ε, Εφευρέτη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, θα είμαστε προσεκτικοί. Είναι και συμβολικό αυτή η επιστολή. Βέβαια είναι συμβολικό γιατί κανείς δεν μας ξέρει, θα πει ποιος μας γράφει. Αλλά θα το στείλουμε και στις μερίδες. Και θα παρακαλέσω κάθε ένα από εσά όπου έχει δυνατότητα να ασχίσει πίεση στην κυβέρνησή του, να τους πει ότι δεν μπορεί την Κυριακή να εκθιάσουν το, την παιδεία και τη Δευτέρα να κάνουν περιορισμός. Μόρτον, πες μας κιόλας κι αν έχεις κάτι για την ε, νεολαία κινή στον προορισμό ή όχι, αλλιώς θα σας κυνηγήσουμε. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξει ξεχωριστή γραμμή για τον προϋπολογισμό στη γνωμοδότηση. Παρανόηση ήταν αυτό. Δεν θα προσθεθεί γραπτή ε, γραμμή για αυτό, αλλά ούτε και για κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω πολλά. Ήταν σαφές το μήνυμα και ήταν και ισχυρό επίσης. Όπως είπε και η Πρόεδρος, πρέπει να υπάρξει κάποια δράση εδώ. Ίσως ε, μια επιστολή προς τα κράτη-μέλη θα ήταν καλή ιδέα κάποιες παρατηρήσεις τώρα στα σχόλια που ακούστηκαν. Ε, η κυρία Φερχόιβεν αναφέρθηκε και στην κατάρτιση δημοσιογράφων. Ξέχασα να τον αναφέρω στην παρουσίασή μου, αλλά αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Δεν βλέπω εκπροσώπους του Συμβουλίου σήμερα, άρα για το Auschwitz θα πρέπει να συζητήσουμε αργότερα και να επανέλθουμε δηλαδή στο θέμα. Θα προσπαθήσω να κανονίσω μια νέα συνάντηση των σχεδόν εισηγητών τέλη Αυγούστου. 31 Αυγούστου, αν μπορείτε. και εκεί θα εξετάσουμε την κατάσταση όπως θα έχει τότε. Το άλλο που μπορώ να πω τώρα είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι λάβαμε ένα σαφές μήνυμα από την Επιτροπή σήμερα. Ωραία, θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την θλιβερή συζήτηση. Α, προθεσμία της τις 31 Ιουλίου. Ωραία. 23 Ιουλίου, συγγνώμη, 23 Ιουλίου για τις ε, τροπολογίες. Σημείο 9. Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Η κυρία Κάμερα δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά το θλιβερό κεφάλαιο του προπολισμού περνάμε σε ένα άλλο θλιβερό θέμα για την ε, Ευρώπη η λεγόμενη πρόταση οδηγία Μάλστρομ για τον περιορισμό της παιδικής πορνογραφία. Θα ήθελα να σα πω με δύο λόγια ποιε είναι οι σημαντικές τροπολογίες που έχω ε, την πρόθεση να υποβάλω στη γνωμοδότησή μου. Πρώτον, προτείνω να μην έχουμε έναν ορισμό του τι είναι παιδί ή παιδική πορνογραφία, γιατί παιδί σε πολλές χώρες είναι ένας ορισμένος όρος. Παραδείγματο χάρη στην ε, Γερμανία, παιδιά είναι άτομα 114 ετών. Η πρώτη οδηγία της κυρίας Μάλστρομ προβλέπει ότι παιδιά είναι άτομα κάτω των 18 ετών. Δεν έχει νομίζω νόημα να έχουμε εδώ μια τέτοια παρέμβαση στην, στα κρατικά θέματα γιατί εάν πούμε ότι είναι όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών θα, τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών θα υπάρχουν προβλήματα σε κράτη-μέλη. Γι' αυτό εγώ προτείνω να λέμε άτομα κάτω των 18 ετών για να μην χρειαστεί να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ορισμό του τι είναι παιδί και τι όχι. Το ίδιο ισχύει και για την παιδική πορνογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρη η πρόταση. Από μια μεριά προσπαθούν να υπάρχουν μια, ένα σαφή ορισμό, από την άλλη μεριά ε, βλέπουμε ότι ο ορισμός αυτός ε, σε ευρωπαϊκή επικράτεια είναι πολύ διαφορετικός. Και βλέπουμε ότι καμιά φορά το να λέμε παιδική πορνογραφία ε, δίνει το συνέστημα ότι είναι κάτι που δεν είναι και πολύ αυστηρό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει οι κολάσιμες πράξεις που αναφέρονται εδώ θα πρέπει να αναφέρονται πολύ σαφώς, δηλαδή σεξουαλικές πράξεις με άτομα κάτω των 18 ετών. Η επόμενη πρόταση να μην υπάρχει νομική ευθύνη ε, των ε, νομικών ατόμων που αναφέρονται στο άρθρο 11 και 12. Δεν καταλαβαίνω κατά πόσον αυτό μπορεί να βοηθήσει ε, την οδηγία. Γιατί ε, κάτι τέτοιο δεν γίνεται οργανωμένο. Δηλαδή, εάν σε μία ένωση νέων γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα μεμονωμένο άτομο που εκμεταλλεύεται τις δομές και γι' αυτό δεν είναι σωστό να αναφερόμαστε σε ε, ενώσεις νέων σχολεία ή άλλες οργανώσεις και να θεωρούμε ότι η δίωξη θα πρέπει να γίνεται στο σύνολο του νομικού προσώπου αυτού, ενώ υπάρχουν μεμονωμένα άτομα που έχουν δράσει. Στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτή η έννοια της ευθύνη νομικών προσώπων και θα πρέπει να το έχουμε ούτε εδώ νομίζω. Το τρίτο σημείο είναι το θέμα της δίωξης σε περίπτωση ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Είχαμε συζητήσει το θέμα χθες, είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο άρθρο 15 παράγραφος 2 όπως αναφέρεται αυτή τη στιγμή στην οδηγία θα πρέπει να απορριφθεί γιατί έτσι τα θύματα ευδερίνονται επιπλέον γιατί θα τους ζητούνται στοιχεία για άτομα που γνωρίζουν τι γίνει. Επιβαρύνεται λοιπόν ο νέος ή το παιδί εάν του λέμε ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει τι έχει γίνει και ιδίως αν πρόκειται για συγγενείς ή γονείς αυτό είναι μια συμπληρωματική επιβάρυνση. Γιατί αυτό θα είναι αντίθετο και με τις, με τις προσπάθειες συγγνώμη, προστασίας του θύματος νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή θέση ώστε αφενός να πούμε ότι βέβαια υπάρχει ευθύνη της κοινωνίας και θα πρέπει να δράσουμε όπου υπάρχουν υποψίες. Από την αμεριά όμως θέλουμε να προστατεύσουμε τα θύματα και να μην τους ασκήσουμε συμπληρωματική πίεση και να μην φέρουμε και τις ομάδες προστασία των θυμάτων σε κατάσταση ε, που να μην θεωρούνται αξιόπιστες. Επίσης προτείνω όσον αφορά ε, την, ε, το ύψος των κυρώσεων να μην γίνεται καμία αναφορά στην ε, οδηγία. Μου φαίνεται ότι δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να ορίσουμε ελάχιστες κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αυτό θα παρενέβαινε σημαντικό στο, στην ομολογία των κρατών μελών. Γιατί θα πρέπει στις ε, πράξεις που είναι φρικτές του άρθρου 3 να υπάρχει χαμηλότερη κύρωση τελικά από εκείνη που προβλέπεται στην ε, η ε, Γερμανία παραδείγματο χάρη για κάτι ίσως λιγότερο σημαντικό. Θα ήταν τελείως παράλογο κάτι τέτοιο. Γιατί εάν ακολουθήσουμε την Κομισιόν θα πρέπει να αλλάξουμε όλο το σύστημα των ποινών στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ενιαίος ορισμός των κορέσιμων πράξεων και από την άλλη μεριά τα κράτη-μέλη θα ορίσουν τις ποινές βάσει του δικού τους δικαίου. Ένα σημαντικό σημείο <clears throat> είναι ότι η πρόταση μετά το άρθρο 13, 13 20 αναφέρεται σε δυνατότητες προστασίας των θυμάτων. Είναι λογικό αυτό. Um- Ίσως όμως δεν είναι επαρκές ιδίω η σκέψη τη πρόληψη θα πρέπει να συμπεριληφθεί περισσότερο στην πρόταση τη οδηγία. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά το να μάθουν οι νέοι πώς μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν το την, την, την επίθεση στο διαδίκτυο. Οι γονεί θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν αυτό. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, ότι μου... Πώς θα πρέπει να συμπεριφερθώ εάν αντιμετωπίσω έναν επιδεξί όταν ήμουν ένα μικρό κορίτσι. Το θυμάμαι ακόμα που μου το είχε πει η μητέρα μου και μου είχε μάθει τι πρέπει να κάνω. θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά λοιπόν σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα που υπάρχουν στο διαδίκτυο να ξέρουν ποιο είναι ο κίνδυνο αν δώσουν τα προσωπικά του στοιχεία. Θα υποβάλω εγώ μια σχετική τροπολογία πάνω σε αυτό και περιμένω να ακούσω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις γιατί νομίζω το θέμα της πρόληψης θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Έκτο και τελευταίο σημείο. που οδήγησε σε πολλές συζητήσεις και στα κρατημέλη και εδώ στο Κοινοβούλιο είναι το θέμα της, ε, της εισαγωγής σε όλη την Ευρώπη ε, προγραμμάτων φραγής. Εγώ είμαι κατά αυτό, γιατί ε, η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται δεν μου φαίνεται ότι είναι σωστή, γιατί ξέρω ότι πολλές αντιδράσεις υπάρχουν έντονες, υπάρχει διαγραφή και λέγεται ότι η φραγή είναι καλή όπου δεν γίνεται η διαγραφή, αλλά εγώ νομίζω ότι η διαγραφή γίνεται πάρα πολύ γλίγορα εάν υπάρχει παρέμβαση παραδείγματος του δικαστηρίου. Το παραγωγμένο υλικό υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν έχει εξαφανιστεί, απλώς δεν είναι εύκολα προσιτό εάν υπάρχει φραγή. Ε, η φρεγή όμως προϋποθέτει μία ε, υποδομή που θα μπορούσε πάντα να χρησιμοποιηθεί για ε, λογοκρισία. Και νομίζω θα ήταν πολύ υπερβολική αντίδραση αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βρούμε ένα λογικό σύστημα αφενός για να προστατεύσουμε τα παιδιά, να υπάρχει δίωξη διεθνώς, διεθνής δηλαδή συνεργασία στην καταπολέμηση των σεξουαλικών πράξεων με άτομα κάτω το 16 αλλά μία ένας περιορισμός της επικοινωνίας και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υποδομής λογοκρισίας δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστή. Θα πρέπει να φροντίσουμε το διαδίκτυο να, είναι, να έχει χέρι τόση εμπιστοσύνης που να παραμένει ένα ε, μέσο ε, επικοινωνίας. Εάν κάποιες χώρες θέλουν να έχουν συστήματα φραγής, ε, δεν μπορώ να τις παρεποδίσω, αλλά δεν θέλω να υπάρχει ε, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο λογοκρισίας. Να υπάρχει απαγόρευση περιεχομένου, να υπάρχει διαγραφή περιεχομένου, αυτό οπωσδήποτε. Αλλά ε, νομίζω το θέμα της φραγής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέμα βασική συζήτηση που κάνουμε και σε άλλους τομείς. Αυτά καταρχήν θα περιμένουμε χαρά να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και ελπίζω από κοινού να μπορέσουμε η πρόταση αυτή οδηγίας να ε, δρομολογηθεί σωστά και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε η παιδική πορνογραφία να καταπολεμηθεί πολύ καλύτερα στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κανέβερ. Έχουν ζητήσει το λόγο ε, διάφοροι συνάδελφοι. Κύριε Φεχάιν, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την, την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία γιατί όχι μόνο χθε, αλλά και προηγουμένω είχαμε πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων. Ακόμα και αν υπάρχουν σε ορισμένα σημεία διαφορές ε, στι απόψεις μα όπω είπε και η κυρία Κάμερεβερτ. Η έκθεση αναφέρεται σε πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Υπάρχουν και διάφορα συμπληρωματικά θέματα που θα μπορέσει να τονίσουμε. Το είπε και η κυρία Καμερεβέρτ, είναι το θέμα της πρόληψη. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της ε, ενημέρωσης των νέων αλλά και των γονιών που δεν ξέρουν το διαδίκτυο, δεν ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι και γι' αυτό δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά του τι οδηγίε του τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς το θέμα της πρόληψης δεν αναφέρεται απαρκώς στην πρόταση της κυρίας Μάλστρομ, ακριβώς επειδή λέει ότι αυτό είναι θέμα των κρατών μελών, αλλά εγώ πιστεύω θα πρέπει να το ζητήσουμε, να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα μέτρα από τα κράτη-μέλη για τον τομέα αυτό. Ένα, Ένα δεύτερο σημείο είναι το θέμα του ορισμού του τι είναι παιδί, γιατί στα διάφορα κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ διαφορετικές έννοιες στη μια χώρα το παιδί είναι μέχρι τα 12, μέχρι τα 14, μέχρι τα 16 και άμα μιλάμε για παιδί είναι πολύ δύσκολο να έχουμε κάτι το ενιαίο σαν αποτέλεσμα. Και μια που στο προήμιο λέμε ότι παιδί εννοεί όλοι που είναι κάτω των 18 μπορούμε αυτό να το αναφέρουμε παντού. Γιατί αλλιώς τα διάφορα ποινικά συστήματα ε, ποινές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού που είναι το θύμα. Ένα άλλο σημείο σημαντικό και που συμμερίζομαι είναι το θέμα των ποινών. Αλλά μου φαίνεται σημαντικό να μην διαγράψουμε απλώς αυτά τα σημεία, αλλά απλώς να πούμε ρητά στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη μέσα στα ποινικά του συστήματα το πόσο σημαντική είναι αυτή η ποινή. Δηλαδή ε, βλέπω ότι πολλές φορές στη χώρα μου ε, δίνεται αναστολή στις ε, κυρώσεις, στις ποινές αυτές και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για ποινή λοιπόν αν δίνεται αναστολή θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη το πόσο σοβαρή και απεχθέα ήταν η πράξη. Ένα άλλο σημείο που συζητιέται είναι το θέμα της ανεμπρόσης των εικόνων στο διαδίκτυο. Γιατί από μια μεριά έχουμε τις σελίδες web, στις σελίδες που μπορεί κανένας να τις βρει παντού, αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό της ε, πορνογραφίας που υπάρχει στο διαδίκτυο. Ε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι σε διάφορου χώρου chat και άλλα διάφορα κλειστά συστήματα, όπου μπαίνει κανένα να το πούμε έτσι με πρόσκληση. Πρέπει δηλαδή κάπως να διαθέσει υλικό για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο ε, υλικό και μία φραγή δεν έχει εδώ απαραίτητο αποτέλεσμα. Γι' αυτό μου φαίνεται ότι το σύστημα της φραγής έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διαγράφονται αυτά τα περιεχόμενα είναι εξίσου γλίγορη αντίδραση όπως μια φραγή. Γιατί παραμένουν αν υπάρχουν κάποιες σελίδες οι οποίες ε, ερευνούν ε, ε, τραπεζικά στοιχεία, σε δύο ώρες μπορούν να εξαφανιστούν από το διαδίκτυο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με αυτά τα πορνογραφικού περιεχομένου ε, chat κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε δομέ, υποδομές που να υπάρχει γρήγορη πρόσβαση ούτως ώστε σε όλη την Ευρώπη να μπορεί να διαγραφεί άπαξ διαπαντός ε, το περιεχόμενο και όχι με μια φραγή. Ο γιος μου μου λέει ότι μια φραγή τη <laughs> ξεπερνάει με... σε λίγα λεπτά. Δεν υπάρχει απόλυτη δηλαδή ε, προστασία με τη φραγή Και αν η νομοθεσία προβλέπει η φραγή να είναι η τελευταία λέξη, υπάρχουν, θα υπάρχουν προσπάθειες ούτως ώστε η πρόληψη και η ε, διαγραφή παραδείγματο να μην έχουν την κύρια προτεραιότητα. Ε, αυτά θα πρέπει να έχουν την κύρια διαγραφή και εκεί που δεν μπορώ να διαγράψω και που δεν πετυχαίνουμε πολλά με ε, πρόληψη και προστασία κλπ. Αν υπάρχουν δηλαδή αυτά σε χώρες όπου δεν έχουμε πρόσβαση, θα πρέπει τα κρατη να δουν τι θα κάνουν βάσει των διατάξεων όμως για την προστασία των δεδομένων. Όπως υπάρχουν και σε πρώτες κυρίες Μάλστρομ. Ένα άλλο σημείο είναι οι ίδιες προσπάθειες που είχαμε και στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ για την συμφωνία SWIFT. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε τη ΣΥΠΑ όσον αφορά τη διαγραφή της παρουσίας της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Γιατί πολύ από το ολικό υπάρχει στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή και θα πρέπει και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δράσουμε. Κατά τα άλλα, με λίγες προσθήκες, που έχουν ήδη συζητηθεί. Μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε με την έκθεση αυτή. Κοιτάξτε, θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Κομισιόν, ε, να προσέξει τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σας άκουσε η Κομισιόν, όπως πρέπει. Ο κύριος Κορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο πριν από μένα και ε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνώ με το ζήτημα του ορισμού για όλους αυτούς τους λόγους που ήδη αναπτύχθηκαν. Γιατί μερικές φορές πράγματι υπάρχει μεγάλη διαφορά στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον, τον όρο ανήλικος. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μεγάλη ε, προσπάθεια σε επίπεδο πρόληψης είναι πολύ σημαντικό για το θέμα αυτό και ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο και τις ε, δυνατότητες συνδρομής ε, προς τα θύματα και αρρωγής ε, των θυμάτων. Νομίζω όμως ταυτόχρονα ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε σαφώς ότι ο βασικός στόχος είναι πάντα η εξάλληψη κάθε πορνογραφικού υλικού. Και αυτό είναι ουσιαστική επιδικής ε, παιδικού πορτογραφικού. Ε, και αυτό είναι ουσιαστική σημασία. Όσον αφορά τη φραγή, η φραγή ε, είναι προσωρινό μέτρο και απευθύνεται κυρίως στις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί όπου είναι πιο πολύπλοκη η δική μας η παρέμβαση. Και κυρίως Κυρίως ε, μιλάμε για τις περιπτώσεις όπου ε, πρόκειται για κράτη, για κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαφορετικό από το θέμα της λογοκρισίας. Είναι, είναι, ένας, ε, ε, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει. Περιορισμός της προσωπική ελευθερία, βεβαίω. Τώρα δεν θέλω εδώ να επισέλθω σε μια φιλοσοφική συζήτηση, αλλά η ελευθερία δεν σημαίνει ε, να δρά κανεί ανεξέλεκτα. είναι φιλοσοφική συζήτηση, έχουν τοποθετηθεί διανοούμενοι φιλόσοφοι. Εδώ μιλάμε για ε, καταστάσεις, έτσι. Άρα, απομάκρυνση εικόνα. Η φραγή δεν είναι μοναδική λύση. Η φραγή ε, είναι μέτρο σε περιπτώσεις που είναι αδύνατο ε, να παρέμβει κανεί. Κυρίως όταν μιλάμε για περιοχές εκτός τη επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να ε, γίνονται ανθρωποκτονίες, δυσάρεστες καταστάσεις, έτσι. Αλλά επειδή εξακολουθούν να γίνονται ανθρωποκτονίε, δεν θα πει ότι εμεί, ε, για παράδειγμα, δεν έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Άρα πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μα απέναντι σε πάση ε, φύσεω αδίκημα. Ε, φραγή λοιπόν εκεί όπου δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πρόληψη και αρρωγή προ τα θύματα. Και θέματα, αυτά είναι δύο θέματα που επίση πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είχε απογορευτεί ό,τι μπορούσε να απογορευτεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι απογορεύσει αυτέ δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Σα το λέω εισαγωγικά. Γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Καμερεβέρ και όσον αφορά το διαδίκτυο. Στη Γερμανία έχουμε μια πολύ ακριβή νομοθεσία στον τομέα αυτό που τελειοποιείται συνεχώς. Και αυτό λύνει το πρόβλημα της κακοποίησης των παιδιών. Εγώ έχω την εντύπωση ότι των αντίον, όσο βελτιώνεται η νομοθεσία, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι ε, κακοποίησεις αυτές. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε μία μελέτη για να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα νομοθετικά μέτρα. Γιατί αυτή τη φορά δεν μπορούμε να πούμε πόσο αποτελεσματικά είναι η νομοθεσία, γιατί μόλις τώρα μαθαίνουμε πολλά πράγματα του παρελθόντος. Και υπάρχουν ε, πολλές άγνωστες περιπτώσεις. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Παραδείγματο χάρη, αν είχε γίνει κάποια κακοποίηση, κάποια σεξουαλική εκμετάλλευση στο παρελθόν, τότε ήταν αυτό απογορευμένο, δεν ήταν, πια ήταν η νομοθεσία που ίσχυε, ποιε ήταν οι ποινέ κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε μία μελέτη, να δούμε κατά πόσο να αυστηρή νομοθεσία βοήθησε ή δεν βοήθησε. Ευχαριστώ κύριε Ρένα. Εγώ θα πάρω το λόγο ως ε, ε, δικηγόρος, σαν δικηγόρος και να πω ότι πρέπει να δούμε πραγματικά πόσο σημαντικά στο ποινικό δίκαιο είναι αυτά και πραγματικά δεν θα προστατήσουμε ιδιαίτερα τα θύματα εάν εγκληματοποιήσουμε περισσότερο. Είναι δύσκολο να πούμε τι πρόθεση είχε ένας θείος που τηλεφώνησε για να πει ότι κάτι είχε γίνει λοιπά. Δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας μετά και το αποτέλεσμα είναι ότι αθωώνεται ε, το εν άτομο. Αυτό δεν είναι όμως υπέρ της ε, προστασίας των ε, θυμάτων. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει να παρέμβουμε στη, στο δικαστικό τομέα. και φαίνεται ότι οι κατάλογοι των ποινών προσαρμόζονται ετήσια στα κρατη Στην Αυστρία μόλις έγινε και είχαμε στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις ε, τέτοιων πράξεων στο εκκλησιαστικό και στον ε, σχολικό τομέα και δεν επιτρέπεται να έχουμε εδώ μία πληθώρα διαφορετικών ε, ποινών, πράγμα που δεν βοηθά το θέμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές υπάρχουν, υπάρχουν αυτές οι, ε, οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιος ε, προσπαθεί να κατηγορήσει παραδείγματο χάρη σε περίπτωση διαζυγίου, χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό άτομα και λόγω του τύπου και του ΜΜΕ υποφέρουν ολόκληρε οικογένειε. Ευχαριστώ κυρία Πινταναλόβα. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι παραμένω αρκετά νέα, αλλά μετά βλέπω και 12χρονα παιδιά με τρομερές εμπειρίες ε, σεξουαλικές, οπότε δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσα θύματα. Βλέπουμε σήμερα ακόμη και παιδιά 6 χρονών να περνάνε πολλές ώρες στο ίντερνετ. Ένας τόσο ξέρει τι βλέπουν εκεί. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουν τα κράτη-μέλη τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο ήδη από την πρώτη δημοτικού γιατί βλέπουν τα παιδιά τέτοιου είδους εικόνε, οπότε πρέπει να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Ευχαριστώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τα παιδιά και τα θύματα. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως η πρόληψη της κακοποίησης είναι ένα θέμα κλειδί, αλλά το ίδιο είναι και το μπλοκάρισμα της αγοράς τέτοιων εικονών. Η διαγραφή είναι μια καλή λύση, αλλά δεν μπορούμε να το επιτύχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο είδους ε, μπλοκάρισμα που χρησιμοποιούμε προαιρετικά στο Αναμένο Βασίλειο για να μπορούμε να έχουμε κάποια πρόληψη μέχρι να γίνει η διαγραφή ελπίζοντας ότι θα γίνει γρήγορα η διαγραφή γιατί όσο παραμένουν κάπου οι εικόνες τόσο ουσιαστικά συνεχίζεται η κακοποίηση του παιδιού. Τώρα όσον αφορά την ηθικολογία. Μπορεί να υπάρχει ηθικολογία, αλλά από την άλλη πλευρά θέλουμε προστασία και αυτό σημαίνει και προστασία δεδομένων και ανωνυμία που είναι σημαντικά. Τώρα όσον αφορά τις καταδίκες, αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά βλέπω εδώ στη διατύπωση να μιλάτε για μέγιστες ποινές δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ορολογία. Δεν μπορώ να πάω εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε ότι υπάρχουν μέγιστες ποινές. Ευχαριστώ κυρία Χάνιμπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, το θέμα μας είναι τα θύματα, το είπαν όλοι. Και βεβαίως το σημείο εκκίνησης είναι η πρόληψη. Αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε. Όμως δεν λειτουργεί πάντα η πρόληψη. Υπήρξαν πολλά προληπτικά μέτρα στο παρελθόν που προφανώς δεν δούλεψαν. Δεν είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ με τον κύριο Μπίσκε ότι αυξάνεται ο αριθμός των κακοποιημένων παιδιών. Νομίζω ότι το ακούμε περισσότερο, αλλά και αυτό είναι καλό, γιατί έτσι μαθαίνουμε να το αντιμετωπίζουμε το θέμα. Υπάρχουν ε, διαφορές ε, απόψεων ε, για το τι πρέπει να κάνουμε, για τη χρήση του ίντερνετ, για τη χρήση μπλοκαρίσματος και γνωρίζω ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και σε άλλες επιτροπές που αφορούν άλλους τρόπους χρήσης του ίντερνετ. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Όπως είπε η κυρία Μαλ Κλάρκιν, στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούμε και το μπλοκάρισμα και την διαγραφή και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα παιδιά θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικό. Τώρα θα συμφωνήσω όσον αφορά τις ποινές. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να πούμε στα κράτη-μέλη τι καταδίκες θα δίνουν. Τίθεται θέμα επικουρικότητας εδώ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες εδώ. Επαναλαμβάνω όμως πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι το βασικό θέμα είναι τα θύματα, τα παιδιά. Ευχαριστώ κυρία Κασιέ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή, με, ε, με την εισηγήτρια όσον αφορά το σύνολο των θεμάτων αυτών και όσον αφορά το θέμα της αναποτελεσματικότητας φραγής. Πράγματι υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη φραγή. Όσον αφορά την ανάγκη σεβασμού, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια το ζήτημα αυτό, Σεβασμό κατά κάποιο τρόπο τη επικουρικότητα των κρατών μελών έναντι του ποινικού του δικαίου. Να επιμείνω κυρίω στο ζήτημα της εκπαίδευση, της ε, ε, πρόληψης μέσω της ε, εκπαίδευση. Μιλάμε συχνά για του γονεί, αλλά συνήθως όσον αφορά το διαδίκτυο, τα παιδιά είναι εκείνα που εξηγούν στου γονεί για τη χρήση του διαδικτύου. Αναφέρεται λοιπόν πολύ ο, ο ρόλο του σχολείου. Λέμε όλοι ότι το σχολείο πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά για να έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία. Αλλά μέσα στο θέμα αυτό τη πρόσβαση τη νέα τεχνολογία από το σχολείο, το ζήτημα αυτό είναι ουσιώδου σημασία. Γιατί διαμέσου του σχολείου ε, θα φτάσουμε στο μέγιστο αριθμό των παιδιών. Και ω το τον πιο νωρί. Γιατί μιλούν μεταξύ του τα παιδιά, συνεργάζονται, μειούν το ένα το άλλο στο διαδίκτυο και καταλαβαίνετε, ε, αν δεν ε, ε, τα έχουμε προειδοποιήσει, εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ζήτημα αυτό. Και συμφωνώ και πολύ ευχαρίστω. Συμφωνώ με την κυρία Νεβεντάλοβα για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εκπαίδευσης, της σύνδεσης με τις νέες τεχνολογίες και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Γιατί βεβαίως τα αισθητήματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ευχαριστώ κυρία Μπερζά κύριος Μάτουλα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ε, σας, εκφράσω κάποιες σκέψεις, όχι μόνο για το θέμα της, της έκθεσης αυτής, αλλά και για την προηγούμενη έκθεση και για πολλές άλλες εκθέσεις. Εδώ μιλάμε για ε, τη σχέση του παιδιού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κοιτάξτε, να σα πω ότι τα παιδιά μα δεν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τι επιπτώσει των υπολογιστών στη ζωή μα, τι επιπτώσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη ζωή των παιδιών μα. Και εκφράζω τώρα και την πικρία μου για τις μειώσεις στο θέμα του αθλητισμού, για παράδειγμα. Και σας λέω το εξής τα παιδιά περνούν, ξεκολουθούν να περνούν πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή τους. Το 1 τρίτο των παιδιών είναι παχύσαρκα. Και με τρομάζει η σκέψη. Σκέφτομαι το μέλλον και σκέφτομαι τι θα συμβεί σε 15 χρόνια ή σε 50 χρόνια. Δεν θα πρέπει να δούμε Πώ προσεγγίζουμε αυτό το θέμα της ε, εξάρτηση του παιδιού με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κοιτάξτε, μην παρεξηγείτε. Ε, εγώ γνωρίζω για τα θέματα των ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχω διδάξει πληροφορική, δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ε, και άλλα ζητήματα και να καταλήξουμε σε κάποιε ιδέε. Όπω για παράδειγμα, να σα πω το εξή. αν δεν έχουμε χρήματα για τον, για τον αθλητισμό, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε στα σχολεία, στο μάθημα της γυμναστικής. Να, να βάλουμε το εξάφλημα, αν θέλετε. Να τρέξουν τα παιδιά με τον υπο... κρατώντα τον υπολογιστή στα χέρια τους. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ένα μήνυμα για το ε, ε, ε τι ε, σημασία έχει ο υπολογιστή στη ζωή του παιδιού. Και τι πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εργασία Τη εισηγήτριας. Στην έκθεση αυτή που αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Σε όσα υπόθηκαν θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Πλέον είναι τόσο έντονη η πληροφορία που λαμβάνουν τα παιδιά, οι νέοι μέχρι 18 ετών, όπως αναγράφουμε στην έκθεση, που είναι δεδομένο πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ότι το παιδί εκείνο, ο νέος εκείνος που θέλει να έχει πρόσβαση σε τέτοιο υλικό θα τη βρει την πρόσβαση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την πρόσβαση σε κάποια τέτοια πηγή τέτοιων στοιχείων. Επομένως πρέπει να δούμε πώς το διαχειριζόμαστε και σωστά αυτό κάνουμε στην έκθεση. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής πρέπει να, καταλάβουμε ότι πολλές φορές αυτές τις πληροφορίες τα νέα παιδιά τις αναζητούν σε κάποιο σημείο μόνοι τους, σε κάποιο σημείο όταν είναι στο σπίτι τους και ε, με κάποιο τρόπο έτσι ε, συνήθως όχι μπροστά σε όλους, όχι μπροστά ε, στους καθηγητές τους, όχι μπροστά στην τάξη τους, ενδεχομένως με κάποιους φίλους τους ή στο σπίτι τους. Άρα είναι εξαιρετικά κρίσιμος ο ρόλος των γονέων εξαιρετικά κρίσιμος. Και δυστυχώς οι γονείς πολλές φορές, ακόμη κι αν μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στον υπολογιστή, αν, μπει στον υπολογιστή ο, γονέας, δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν έχει τη γνώση. Γιατί ε, δυστυχώς η διαφορά ε, στην αντίληψη για τα πράγματα αυτά, ειδικά με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη παραμένει αυτό το χάσμα μεγάλο και έχουμε χρέος ειδικά στο πεδίο αυτό της ενημέρωσης των γονέων για τους κινδύνους, να έχουμε ακόμη πιο έντονες προσπάθειες στη συνέχεια. Ich möchte das Θα ήθελα να υποστηρίξω ακριβώς αυτό που είπατε. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό που είναι σημαντικό είναι να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, να έχουμε σχολεία γονέων αν θέλετε. Δηλαδή οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι αν δεν ενδιαφερθούν είναι συνυπεύθυνοι. Δεν μπορούμε να αναθέσουμε την ευθύνη αυτή στα σχολεία ή τουλάχιστον θα πρέπει και να έχουμε τη διτή προσέγγιση και οι γονείς και τα σχολεία. Θα αναφερθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν σε αυτό που είπε ο κύριος Μπίσκι είναι ουσιαστικό σημείο γιατί είχαμε και μια ακρόαση και είχα συζητήσει και με πολλούς ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σαφείς αναλύσεις ή μελέτες όσον αφορά τον αριθμό των υποθέσεων, την εξέλιξη κλπ. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά ένα παράδειγμα από την Αγγλία. Είπανε ότι μέσω της φραγής παρεμποδίστηκαν 20 ή 50.000 ε, προσεγγίσεις του θέματος αυτό. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, συστήματα αυτόματης προσέγγισης και ξέρουμε ότι αυτά τα άτομα ε, κάθε 5 λεπτά περίπου μπορούν να εξετάσουν αυτόματα κατά πόσον έχει, είναι φραγμένη η σελίδα, η εικόνα που έχουν βάλει στο διαδίκτυο και αν είναι φραγμένη την ξαναβάζουν κάπου αλλού. Αμέσως. Λοιπόν, θα πρέπει να είχαμε συγκεκριμένες μελέτες γιατί νομίζω ότι μια καλή, σωστή ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη όλων των στοιχείων και με συνεργασία της Ευρωπόλ και άλλων που γνωρίζουν την, ε, το περιβάλλον αυτών θα μπορέσουμε να ξέρουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων. Okay. Jetzt kommt die Πρόεδρος, πολύ ωραία. Η Κομισιόν τώρα. Ο κύριος Σέζαρ Αλόνσο Ρεάτρε. Παρακαλώ. Ε, thank you very much. Ε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Γιάκουμ Μπορατίνσκι, επικεφαλές του τμήματος καταπολέμησης οργανωμένων κλίματων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία, γι' αυτό ήρθαμε όλοι σήμερα εδώ. Πρόκειται για ε, μία από τις πρώτες προτάσεις ε, επί της ποινική νομοθεσίας ε, που έχει προτείνει η Κομισιόν επί συνθήκης της Λισαβόνας με το Κοινοβούλιο σε ισότιμη θέση ως νομοθέτης με το Συμβούλιο. Οπότε παρακολουθούμε πολύ τη διαδικασία και γενικά θεωρούμε ότι η ποιότητα της πρότασης θα βελτιωθεί εξαιτίας αυτής της νέας πλήρους νομοθετικής διαδικασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα περνάω στην ουσία. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση Ίσως δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλα, αλλά θα επικεντρωθώ στα σημαντικά. Καταρχάς, να θυμάστε ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στο θέμα της φραγής. Είναι και νέο θέμα. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια συνολική προσέγγιση στο θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών με μέτρα που αφορούν την δίωξη, μέτρα που αφορούν την ε, συνδρομή των θυμάτων και τέλος ε, και με θέματα που αφορούν την πρόληψη, όπου θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Επίσης, κάτι άλλο που αποτελεί ιδιαιτερότητα αυτών των εγκλημάτων είναι ο σημαντικός ρόλος ε, του ίντερνετ και γενικά της ε, ηλεκτρονικής πρόσβασης. Γενικά, πολλοί έχουν επιστήσει την προσοχή στον ρόλο του ίντερνετ, αλλά παρακαλώ ας θυμάστε ότι αυτή η πρόταση είναι πολύ πιο συνολική. Καταρχάς, υπάρχει μία βασική δήλωση όσον αφορά τον όρο παιδική πορνογραφία. Καταρχάς αναρωτιόμαστε αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο, γιατί αυτή η παιδική πορνογραφία δεν έχει καμία σχέση με την πορνογραφία. Μιλάμε για κατάπτυστη κακοποίηση των παιδιών εδώ. Αυτό είναι η παιδική πορνογραφία. Παρόλα αυτά, επειδή χρησιμοποιείται και σε διεθνής, ε, στο διεθνές περιεχόμενο, χρησιμοποίησαμε τον όρο παιδική πορνογραφία παρόλο που πλέον ε, κερδίζει έδαφος και ο όρος ε, εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Να πω ότι σε μία έκθεση μη κυβερνητικού οργανισμού ανέφερε ότι 44% αυτών των εικόνων περιείχαν βιασμούς ή βασανιστήρια. Μεγάλο ποσοστό αφορούσε παιδιά κάτω των 10 ετών. 23% ε, αφορούσε παιδιά κάτω των 6 ετών. Ας τα θυμόμαστε αυτά τα νούμερα όταν μιλάμε για παιδική πορνογραφία. Τώρα, για τη φραγή. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε φραγή. Για να καταπολεμήσουμε την παρουσία αυτών των εικόνων στο διαδίκτυο χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες. Μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε αρκετή επιτυχία στο να διασφαλίσουμε ότι όταν δημιουργείται μια ιστοσελίδα με τέτοιες εικόνες η απάντηση από τους παρόχους του διαδικτύου και τις διοκτικές αρχές είναι αρκετά άμεση και κατεβαίνουν αυτές οι σελίδες αρκετά γρήγορα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ιστοσελίδων στις οποίες έχει πρόσβαση κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοξενούνται σε ιστοσελίδες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς. Συχνά οι διοκτικές αρχές μιλάνε για πιθανή τοποθεσία τους, δεν μπορούν καν να πούν με σαφήνεια ποια είναι αυτή η τοποθεσία. Αν και συχνά βλέπουμε Ρωσία Είπα, Κίνα και άλλες χώρες εκτός ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Υπάρχει κάποια πρόοδο στη συνεργασία μας με αυτές τις χώρες, αλλά δεν είναι επιτυχής προς το παρόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές φορές υπάρχουν ε, ιστοσελίδες που παρόλο που έχει γίνει αναφορά για αυτές, δύο μήνες μετά παραμένουν online. Οπότε, η φραγή θεωρήθηκε από αρκετά κράτη-μέλη ως απαραίτητο συμπληρωματικό τονίζω μέτρο μέχρι την διαγραφή οριστική των εικόνων. Έχει χρησιμοποιηθεί στη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία με επιτυχία προκειμένου να μειωθεί η δυνατότητα πρόσβασης. Τώρα υπάρχουν κάποια επιχειρήματα κατά της φραγής. Θα τα αναφέρω ένα-ένα. Καταρχάς, παραβίαση του, της ελευθερίας του λόγου και των ελευθεριών του ανθρώπου. Όμως είμαστε αρκετά σίγουροι ότι εδώ δεν πρόκειται για ελευθερία λόγου ή ελευθερία πληροφόρησης. Τώρα, ο άλλος φόβος ότι αυτοί οι μηχανισμοί φραγής θα ξεκινήσουν να ισχύουν για εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και μετά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται και για άλλο περιεχόμενο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε η Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τέτοιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες του κόσμου για μείωση της ελευθερίας του λόγου. Έχει επαναληφθεί πολλές φορές αυτή η δήλωση, αποτελεί σαφή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, το άλλο επιχείρημα, ότι είναι πολύ εύκολο να το παρακάμψουμε. Από δείχνει εμπειρία και αυτό το έχουμε δει και στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με την παιδική πορνογραφία δεν γνωρίζουν καλά τους υπολογιστές κάποιοι είναι αλλά οι περισσότεροι όχι και αυτοί που λένε ότι είναι τόσο εύκολο να παρακάμψουν τα εμπόδια ας κάνουμε μια δοκιμή στο μέλλον να δούμε πόσο εύκολο είναι ο συνάδελφος ο Τσεσάρα Αλόνζο δεν είναι ειδικό, αλλά γνωρίζει από οι υπολογιστές και προσπάθησε να καταφέρει να παρακάμψει τους φραγμούς και δεν τα κατάφερε και υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς δεν θα τα καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτές τις φραγές. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να περιοριστούμε η δυνατότητα του να δει κανείς εικόνες κακοποίησης. Είπε ένα συνάδελφό σας ότι κάθε φορά που κάποιος βλέπει μια τέτοια εικόνα, ένα παιδί, ένα πραγματικό παιδί, θυματοποιείται. Και υπάρχει και ένας ρεαλιστικός ε, λόγος ακόμη. Η αστυνομία μας λέει ότι αυτή η φραγμή αποθαρρύνουν τους ε, πιο χλιαρούς εγκληματίες και έτσι παραμένουν ε, αυτή που είναι η πραγματικά επικίνδυνη και μπορεί και η αστυνομία πλέον να επικεντρώνεται στις πιο σημαντικές υποθέσεις. Okay, I think Αρκετά για τη φραγή. Βεβαίως ε, μπορούμε να σας παρέχουμε και περισσότερες πληροφορίες αν τις επιθυμείτε επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η καλύτερη λύση, δεν είναι και η λύση που θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά μπορεί να μειώσει την πρόσβαση σε εικόνες παιδικής πορνογραφίας. Τώρα, ορισμός της παιδικής πορνογραφίας και ορισμός του παιδιού. Εδώ δεν λειτουργούμε εν μέσω καινού έχουμε ως ε, θεμέλιο λίθο τη σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιού που δίνει ορισμό για την ηλικία. Τώρα, όσον αφορά το πώς ορίζουμε την παιδική πορνογραφία, βασιζόμαστε σε πολυετή συζητήσεις ε, ειδικών που οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση επί του θέματος. να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να αλλάζουμε αυτά τα πράγματα όποτε θέλουμε και να θυμόμαστε επίσης ότι η παιδική πορνογραφία και ο ορισμός που δίνουμε λαμβάνει υπόψη όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει. Τώρα, επί να πω ότι ο ορισμός της παιδικής πορνογραφίας δεν πρέπει να περιερίζεται μόνο στις σεξουαλικές πράξεις, δηλαδή στον εξαναγκασμό παιδιών ε, να επιδεικνύουν τα γενετικά τους όργανα ή στις ε, σεξουαλικές δραστηριότητες. Σε αυτό υπάρχει σαφή συνένεση ότι πρέπει να καλύπτονται και άλλες μορφές κακοποίησης. Άλλο ένα θέμα είναι η εικονική παιδική πορνογραφία, δηλαδή εικόνες που έχουν δημιουργηθεί στον υπολογιστή που μοιάζουν με παιδιά αλλά που δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για πραγματικό παιδί που απεικονίζεται αν και ορισμένες φορές ε, μπορεί να έχει γίνει ένα κολάζ έτσι ώστε να υπάρχει από πίσω ένα πραγματικό θύμα αλλά να έχει επεξεργαστεί η εικόνα έτσι ώστε να μην φαίνεται, φαίνονται ακριβώς ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εκεί οι επιστημονικές ερεύνες δείχνουν ότι το να παρακολουθεί κάποιος να βλέπει εικόνες κακοποίησης παιδιών είναι ένα βασικό βήμα στο να περάσει στην ε, κακοποίηση παιδιών στην πραγματική ζωή. Έτσι βλέπουμε ότι 40% των καταναλωτών παιδικής πορνογραφίας έχουν όντως ε, κάνει τέτοιου είδους εγκλήματα στην πραγματική του ζωή. Άρα λοιπόν διευκολύνει η πρόσβαση σε εικόνες της, τα, τα εγκλήματα πραγματικές κακοποίησης. Τώρα όσον αφορά την πρόληψη. Καταρχάς έχουμε μια υποχρέωση έναντι των κρατών μελών να παρέχουμε προγράμματα παρέμβασης για τους ε, σεξουαλικούς εγκληματίες που κάποια στιγμή βγαίνουν από τη φυλακή αλλά μπορούν να παραμείνουν κίνδυνος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα πρόληψης έναντι αυτών των ατόμων. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις φάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν άτομα που έχουν καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα και απαγορεύεται να εργάζονται με παιδιά. Αυτά που θα μπορούν να διαβεβάζονται στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αποφύγουμε την υποτροπή τους. Όμως, επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε με οδηγία για το ποινικό δίκαιο, Υπάρχει και ένα συνάδελφος ο οποίος ασχολείται με το πρόγραμμα της Επιτροπής για ασφαλέστερο ίντερνετ που εδώ και χρόνια προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς ε, να βελτιώσουν την ασφάλεια στο ίντερνετ και έχει δημιουργήσει και ένα δίκτυο τηλεφωνικών γραμμών στα κράτη-μέλη που επιτρέπουν την αντιμετώπιση της κακοποίησης ε, στο διαδίκτυο online. Όλα αυτά είναι βασική κρίκη στην πρόληψη της κακοποίησης, όμως επαναλαμβάνω, σε μια οδηγία ποινικού δικαίου με βάση τη συγκεκριμένη νομική βάση που έχουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ιδιαίτερα, να περάσουμε σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές τις πτυχές. Θα ολοκληρώσω εδώ. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά τη δέσμευσή μας για στενή συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας συγχωρείτε, τη δέσμευσή μας για διάλογο. Θα υπάρξει και η πολύ σημαντική ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέλη Σεπτεμβρίου θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και τα τεχνικά θέματα. Παραμένουμε στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις, θέλετε διευκρινήσεις, γιατί έχετε κάθε δικαίωμα να είστε πλήρως ενημερωμένοι για το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ενημερωτικά όλα αυτά. Ευνόητα. Για εκείνους που δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα τόσο πολύ με το θέμα. Σήμερα αποκτήσαμε νομίζω μια ε, γενική εικόνα όσον αφορά το πολύμορφο των προβλημάτων αυτών. Και όταν λέτε ότι αυτή είναι μια οδηγία που παρεμβαίνει στο ποινικό δίκαιο, πρέπει να σκεφτούμε πού και πότε μπορούμε να εργαστούμε και για την πρόληψη. Και αυτό θα πρέπει να μας το πείτε κάπου, γιατί η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, το είπατε και εσείς. Κάποιος ακόμα από την Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα απαντήσω σήμερα στην πιο πολυχρησιμοποιημένη γλώσσα. Είμαι από τη Γενική Διευθυνσή της Κοινωνικής Πληροφόρησης και των ΜΜΕ. Έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ και 10 χρόνια. Εργαζόμαστε δηλαδή κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Πολλά τροποποιήθηκαν τα 10 τελευταία χρόνια. Το θέμα δηλαδή είναι ένα θέμα που όσο και περισσότερο είναι γνωστό στην κοινή γνώμη. Θα θέλαμε ορισμένα κράτη-μέλη να ε, δεσμευτούν περισσότερο, να οργανωθούν περισσότερο. Έχουμε το πρόβλημα ότι οι οργανώσει με τι οποίε συνεργαζόμαστε σε αυτά τα δίκτυα δεν έχουν συγχρηματοδότηση από τα κράτη και σιγά σιγά προσπαθούν να μαζέψουν τα χρήματα από εδώ και από εκεί και δεν λειτουργεί πάντα το σύστημα σωστά. Δεν επιτρέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, να επιδοτεί αυτές τις δομές επί χρόνια και χρόνια επειδή τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ασχοληθούν. Θα σας πω γιατί Εντάξει, τάξη μεγέθους συζητάμε η InHop θέση συντονισμού αυτών των hotlines όπου μπορούν οι πολίτες να στραφούν έχουμε 100.000 δηλώσεις για, για παιδοφιλία κάθε χρόνο που προωθούν μετά τις αρμόδιες αρχές. Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να διαγράψουμε τα περιχώμενα αυτών των ιστοσελίδων είναι σαν τον αγώνα με τους ανεμόμυλους. Σε χρό... Θα πρέπει να βράσουμε ακόμα πολλά χρόνια κατά μου για να καταφέρουμε αυτού του περιεχόμενου στις λύσεις να διαγράφονται αποτελεσματικά από το διαδίκτυο. Μέχρι στιγμή δεν είναι δυνατόν και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει και η φραγή σαν συμπληρωματικό μέτρο. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παραλυσμό γιατί ο εικονικό κόσμο δεν πρέπει να υπάρχει σε διαφορετικού κανόνε ότι ο πραγματικό, η αστυνομία η οποία όταν πρόκειται για έντυπο υλικό αυτού του τύπου έχει το δικαίωμα να το καταστρέψει. Αλλά αν υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες για να μην έχουμε λογοκρισία. Γιατί αν δεν επιτρέψουμε την πρόσβαση θα είναι λογοκρισία. Λοιπόν μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Θα πρέπει ήδη ίδιοι, ε, οι κανόνες να ισχύουν στο ε, διαδίκτυο όπως και στην πραγματική ζωή. Αυτό δεν αναφέρεται ποτέ όμως. Και μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά το ε, σενιές ελάχιστες ποινές. Ε, σωστά ότι πολλές φορές αυτά τα στοιχεία ανταλλάσσονται σε κλειστά δίκτυα. Είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί και εμάς. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο καταναλωτής στη χώρα Α που ανταλλάσσει με κάποιον στη χώρα Β ε, απειλείται από μια ε, ποινή τριών μηνών στη χώρα Β ο άλλος όμως με ελάχιστο δύο ετών. Είναι περίεργο και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποιες ελάχιστες ποινές για να δείξουμε ότι ακριβώς χρειάζεται να υπάρχει διακανονισμός σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ναι, απαντήσετε εδώ σε διάφορους συναδέλφους. Ξανά θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Um, I'm really sorry because I... Συγγνώμη, γιατί δεν αναφέρθηκα στο θέμα των κυρώσεων ε, στην προηγούμενη μου δήλωση. Πολύ σύντομα να σας πω ότι γιατί ακριβώς ε, καθορίζουμε αυτό το επίπεδο ποινών. Γιατί αυτό ε, μας το επιτρέπει ε, η συνθήκη της Λισαβόνας. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το στάδιο εξέλιξη του, του ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να καθορίσουμε ελάχιστο και μέγιστο όριο να σα το πω, γιατί άκουσα αυτές τις ανησυχίες να εκφράζονται και εδώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν για ένα συγκεκριμένο αδίκημα η οδηγία αναφέρει ε, τουλάχιστον πέντε χρόνια ποινή, τότε το κράτο μέλος στον ε, Εθνικό Ποινικό Κώδικα θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον πέντε χρόνια. Πέντε, έξι, εφτά μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό. Τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή από αυτό το επίπεδο και πάνω. Γιατί το κάνουμε αυτό. Όπω είπε και ο συνάδελφο, είδαμε μεγάλε διαφορέ όσον αφορά το επίπεδο τιμών, ποινών ανάμεσα στα κρατημέλη. Από δύο χρόνια μέχρι 15 χρόνια ε, προβλέπονται ποινέ για ένα συγκεκριμένο δίκημα. Και είναι πολύ σημαντικό να ε, στείλουμε ένα μήνυμα συνέπεια ότι πρόκειται για σοβαρά αδικήματα που ε, πρέπει να τιμωρούνται και πρέπει να απαντά ε, στο επαρκές επίπεδο και ε, το ποινικό δίκαιο. Επίσης, όσον αφορά την ευθύνη των νομικών προσώπων. Δεν λέμε ότι είναι ποινικέ οι ευθύνε αυτέ, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι, όπως και σε πολλά άλλα σημεία, ότι εδώ ε, τα εφιστάμενα μέσα. Αυτό κάνουμε στο παρελθόν και εδώ έχουμε τα διεθνή μέσα δεν αναφέρουμε τις λεπτομέρειες, γιατί πιστεύουμε και αυτό είναι σημαντικό τμήμα μία συνεπούς απάντηση. Γιατί ορισμένες επιχειρήσεις διευκολύνουν ή επιδίδονται σε τέτοια δικήματα. Να σας πω επίσης ότι μία νέα μορφή εγκλήματος που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό το θέμα του, του τουρισμού παιδικής και πορνογραφίας. Και εδώ προσπαθούμε να πιάσουμε και τους ενδιάμεσους που, ε, ε, ε, για να τιμωρηθούν και αυτοί που μεσολαβούν ώστε να γίνονται αυτές οι, να, γίνονται αυτές δραστηριότητες. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια τη ευθύνη των νομικών προσώπων. Ε, Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σα δώσω συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι... Ευχαριστώ. Χρειαζόταν νομίζω να με δώσετε αυτέ τι διευκρινήσει. ρώτησαν η, η κυρία Μακλάκ και μετά η κυρία Καμερέβερ. Ναι. Να το ξεκαθαρίσω. Όταν λέτε όταν μιλάτε για ελάχιστο για μέγιστο, τι εννοείτε. Ότι, ότι πρέπει ε, η ποινή αυτή να, ε, να την εκτίσει κανείς την ποινή του ε, κανονικά, δηλαδή να μην, να μην ε, βγει από τη φυλακή νωρίτερα ή μιλάτε για ελάχιστο και για μέγιστο όριο. Εμεί ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να μελετήσουμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη και πώ ακριβώ εκτείει κανεί την ποινή του. Αλλά αυτό ε, αφορά το σοφρονιστικό σύστημα των κρατών μελών και τι αποφάσει των δικαστηρίων. Υπάρχουν χώρε όπου κανεί ε, μπορεί να βγει με αναστολή. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να εναρμονιστούν τα ζητήματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλά και μόνο μιλάμε για τι διατάξει του κώδικα. Αλλά εσεί χρησιμοποιήσετε και τη λέξη μέγιστο. Ε, ελάχιστο του μέγιστου. Ελάχιστο του μέγιστου. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να το εκφράσω. Αλλά έτσι ε, ε, οικοδομούμε εμεί την ποινική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δύσκολο. Αν πούμε δηλαδή στην οδηγία ποινή τουλάχιστον πέντε χρόνων, γιατί αυτό χρησιμοποιούμε στην οδηγία, Uh, Αυτό σημαίνει ότι στον ποινικό κώδικα της χώρας Α το συγκεκριμένο αδίκημα που αναφέρεται στην οδηγία θα πρέπει να τιμωρείται με μέγιστη ποινή, λέει ο μιλητής, από πέντε χρόνια ή περισσότερο. Εξαρτάται δηλαδή από την εθνική νομοθεσία. 10-15 χρόνια μπορεί να το ξεπεράσει. Αυτό που θέλουμε να πούμε σε τελευταία ανάλυση είναι ότι η ανώτατη ποινή με βάση τον ποινικό κώδικα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το όριο που αναφέρεται στην οδηγία. Λοιπόν, εντάξει. Η κυρία Καμερέβερτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή και υποκοδομητική συζήτηση που είχαμε σήμερα. Έχω να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις με εξέπλησαν οι δηλώσεις Κομισιόν που αφενός λέει ότι ε, θέλουν μια πολύ ευρία προσέγγιση. Απ' την άλλη μεριά για την πρόληψη λένε ότι πρόκειται μόνο για κάποια μέτρα ποινικού δικαίου ε, γιατί νομίζω το θέμα της ε, πρόληψης και συμφωνούμε πάνω σε αυτό όλοι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να αντικατοπτρίστηκε και στην οδηγία. Όσον αφορά τα ύψη των ποινών, θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο χρειάζεται στην Ευρώπη να έχουμε ενιαίο ποινικό δίκαιο. Εάν το κάνουμε όμως αυτό θα πρέπει να το κάνουμε παντού, για όλο το ποινικό δίκαιο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα τομέα, γιατί τότε πραγματικά θα αναμίξουμε τόσο πολύ τα ποινικά συστήματα των κρατών μελών και θα οδηγηθούμε σε πάρα πολλές ασυνέπειες και γι' αυτό ε, ευχαριστώ στην φορά αλλά για αυτά που είπε για άλλη μια φορά και θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε καθόλου το θέμα της αναλογικότητας των μέτρων. Αυτό είναι μια βασική αρχή νομική και της δικαιοσύνης που θα πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση που εξετάζουμε το θέμα κακοποίησης παιδιών. Αυτό που είπε η κυρία Ράινερ λοιπόν μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά και το θέμα της φραγής, μπορούμε να τη ζητήσουμε διαμακρών. Το θέμα που τίθεται όμως δεν είναι ε, ότι πρέπει να υπάρχει ελευθερία επικοινωνία στους εγκληματίες ή η ελευθερία για την παρουσίαση σεξουαλικών πράξεων κατά παιδιών στο διαδίκτυο. Προφανώς είναι κολάσιμες πράξεις αυτές και προφανώς θα πρέπει να προβλέπονται το ποινικό δίκαιο. αλλά αυτό το είπε η κυρία Φεάρεν στην περίπτωση των τραπεζών και αναρωτιόμαστε γιατί λειτουργεί για ε, θέματα οικονομικά το θέμα της διαγραφής και εδώ που πρόκειται μας για παιδιά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, έχει, ότι ό,τι έχει γίνει έχει γίνει όταν φτάσουν οι εικόνες στο διαδίκτυο γιατί δεν μπορούμε λέω, εκεί να αντιδράσουμε εξίσου γρήγορα. Γιατί το θέμα της φραγής δεν είναι μόνο το θέμα της ε, παιδικής ε, πορνογραφίας και κακοποίησης των παιδιών. Είναι ότι για τη φραγή χρειάζομαι μία υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οποιοδήποτε έλεγχο της επικοινωνίας. Δεν εννοώ ότι το θέλω αυτό η Κομισιόν, αλλά το είδαμε στη Γερμανία όταν συζητήσαμε το θέμα ότι μετά εξετάστηκε στους ναι και τι άλλο θα μπορούσαμε να φράξουμε όπου καμιά φορά α, πρόκειται για περιεχόμενο απλώς μη επιθυμητό, όχι ε, διώξιμο. Λοιπόν, θα πρέπει εδώ να αμυνθούμε εκ μιας αρχής. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενδυναμώσουμε τη διεθνή συνεργασία και ακριβώς αυτές οι συμφωνίες που έχουμε και σε άλλους τομείς με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες να τις, ε, να τις εισαγάγουμε και εδώ. Και οι εμπειρίες δείχνουν ότι το περιεχόμενο του διαδικτύου μπορεί να διαγραφεί πάρα πολύ γρήγορα αν το θέλουμε. Οι φρεχές δεν είναι 100% σίγουρες και κατάλογες φραγής θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ε, μια κατάλογο περιεχομένου για εκείνου που θέλουν άμεση πρόσβαση σε αυτά τα, τα θέματα, σε αυτές τις σελίδες. Γιατί το θέμα δεν είναι να καθαρίσουμε, αν θέλετε μόνο το διαδίκτυο από αυτά τα θέματα αλλά και τα δίκτυα peer to peer αυτά δηλαδή που δεν είναι στο δημόσιο τομέα του διαδικτύου και εδώ ο κίνδυνο είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι γενικά στο διαδίκτυο. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου την αλογικότητα των μέτρων και να δούμε κατά πόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε σε όλη την μικρά της Ευρώπης μια τέτοια υποδομή με την οποία μπορούν να γίνουν και πολλά άλλα. Εγώ είμαι απόλυτα αντίθετη με αυτό και θα μου φαίνονταν καλό να λέγαμε ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να παρεμποδίσουμε τι γίνεται στην Αγγλία, στη Σουηδία ή σε άλλε καθολικέ χώρε, αλλά δεν χρειάζεται να το επιβάλλουμε σε όλη την Ευρώπη. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε προχωρήσει. Α, και κάτι άλλο, μην το ξεχάσω, γιατί υπάρχει ένα σφάλμα εδώ που σας κάνει εντύπωση. Η τροπολογία 14 για το άρθρο 2β Υπάρχει ένα τυπογραφικό σφάλμα. Δεν αφαίνεται η εικονική, εικονική ε, σεξουαλική πράξη. Δεν, ήταν, δεν το σκοπεύω να το κάνουμε αυτό. Θα παραμείνει ως έχει. Η μόνη ε, τροπολογία, η μόνη αλλαγή μάλλον είναι το θέμα της, ε, το τα παιδιά ε, από τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 Πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Έχετε χρόνο μέχρι τις 16 Ιουλίου, την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, δηλαδή να υποβάλλετε τροπολογίες. Η συζήτηση θα συνεχιστεί γιατί στις 28 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας αυτό το θέμα. Λοιπόν, τροπολογίες μέχρι την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας και μετά στις 28 Σεπτεμβρίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πολύ καλή εισαγωγή. Ίσως στην αρχή ήμουν πολύ αυστηρή γιατί θεωρούσα ότι δεν ήταν καλό να μιλάτε εκεί μεταξύ σας και εδώ πέρα οι συνάδελφοι να προσπαθούν να παρουσιάσουν την άποψή σας. Εμείς σας ακούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ τους, την Κομισιόν, ευχαριστώ τους συναδέλφους που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν και όλους τους σχιώδες. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης πρωτοβουλία των πολιτών. Και καταρχήν αναρωτήθηκα τι σημαίνει αυτό. Και ομολογώ ότι όταν ασχοληθεί κανένα με το θέμα, βλέπει Τι καταφέραμε με αυτή τη συνθήκη της Όχι μόνο τον ε, ε, πρόεδρο του Συμβουλίου που δεν έχει τίποτα να πει, ε, τη γυριάσωνα που δεν ξέρει τι γίνεται, αλλά και μια πρωτοβουλία των πολιτών που πάλι δεν ξέρει κανένας ποιος είναι πολίτης, ποιος μπορεί να υπογράψει, ποιος ελέγχει κατά πόσο πρόκειται για πολίτες. Δύσκολα τα πράγματα. Θα χρειαστούμε πολύ χρόνο νομίζω να περάσουμε στην πραγματικότητα. Η κυρία ε, Ρόζα Φοντούν έχει το λόγο. Ε, ε, e, Ευχαριστώ, Ντόρις. Θα προετοιμάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μα για αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ 100% με όσα είπατε και εσείς, Πρόεδρε, πριν από λίγο πρωτοβουλία των πολιτών ορίζεται ως μία από τις βασικές καινοτομίες της ε, ε, συνθήκης Λισαβόνας. Αλλά δεν έχει οριστεί με διεξοδικό τρόπο. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο λοιπόν, αλλά και ε, οι υπόλοιποι δεσμεύονται και άλλοι φορείς δεσμεύονται για να εκφράσουμε συγκεκριμένα αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε οι πολίτες να καταλάβουν πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς γίνεται και ε, να μην ε, αισθάνονται απογοητευμένοι όσον αφορά το βαθμό επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφτάνουν ε, χιλιάδες ιδέες, προτάσεις, υποδείξεις. Όσον αφορά τα θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και τώρα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να μην παρεμποδίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες όλες στην πράξη. Να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας κυρίως σε ορισμένα θεμελιώδη θέματα, κεντρική σημασία θέματα. Και υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι περισσότερο φιλοσοφικού χαρακτήρα. Τώρα, πρώτα απ' όλα να δούμε γιατί συμπεριλάβαμε το θέμα αυτό στη συνθήκη, Γιατί εδώ και χρόνια πιστεύουμε ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στου πολίτε και στα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δηλαδή ε, τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούν στον εαυτό του και δεν έχουν καμία επικοινωνία με του πολίτε. Αυτό το χάσμα είναι κατά κάποιο τρόπο ε, θέμα που απασχολεί όλου τα τελευταία χρόνια. Και ακριβώ γι' αυτό ε, υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών. Δηλαδή ε, να συγκεντρώνεται ένα εκατομμύριο υπογραφές, υπήρξε ένα πράσινο βιβλίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήρθε σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το θέμα αυτό της πρωτοβουλία των πολιτών και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Και εδώ θέλω να την προσοχή σας σε, στο πρώτο θέμα, στο οποίο υπάρχουν ορισμένε επιφυλάξεις. Περίπου 300 από τις οργανώσεις αυτές ανταποκρίθηκαν στην ε, έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι αντιπροσωπεύουν όμως αυτές οι οργανώσεις όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες. Αν θέλετε λοιπόν η ενημέρωση γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και υπάρχουν ορισμένοι που δεν γνωρίζουν τίποτα, μα τίποτα απολύτως για το θέμα αυτό. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ε, χρησιμοποίηση των μέσων που υπάρχουν στη διάθεσή μα, πράσινο βιβλίο, ιστοσελίδα κτλ. Ε, υπάρχουν όμω οργανώσει που είναι πολύ καλά οργανωμένε και που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και έχουν ε, μεγάλη δυνατότητα ενημέρωση. Ε, αυτές λοιπόν οι οργανώσεις ε, είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων αυτών. Τώρα πριν φτάσουμε στα θέματα του παραδεκτού κτλ., θα διαβάσετε το έγγραφο. Να σας πω το εξής. Στην Επιτροπή Πολιτισμού εμείς ασχολούμαστε με ανακοινώσεις προς την κοινωνία των πολιτών. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα ενημερώσει τους πολίτες για αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει η πρωτοβουλία των πολιτών. Μα ακριβώ έχουμε αυτές τις οργανώσεις που προσφέρθηκαν. όσον αφορά ακριβώς τη συγκέντρωση των υπογραφών αυτών. Και ε, αν θέλετε, για να καταλάβουν οι άνθρωποι ε, τι ακριβώς δυνατότητες έχουν, γιατί είναι πολλές οι δυνατότητες, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή την απευθύνομαι και στους συναδέλφους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία θα πρέπει να περιέχει το έγγραφο. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο, στο είδος των πληροφοριών. Τι είναι δυνατόν να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κοιτάξτε, δεν θέλουμε να υπάρχουν πολλά σημεία που και στην, και στην, ε, στην να μην γίνεται τίποτα και να απορρίπτονται όλα αυτά. Εμεί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εμπόδια στην πρωτοβουλία των πολιτών. Αντίθετα, θέλουμε να την ενθαρρύνουμε για να συμμετάσχουν, ε, για να υπάρχει όσο περισσότερη ενεργό συμμετοχή στην νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο ασχοληθεί με αυτέ τι πληροφορίε. Σα είπα ότι πρέπει να ασχοληθούμε ε, με το αποκεντρωμένο επίπεδο. Εκεί δηλαδή όπου μπορεί να βρει του αρμόδιου ο πολίτη. Ε, πολλά ερωτηματικά λοιπόν υπάρχουν όσον αφορά αυτή την πρωτοβουλία μπορεί να φαίνεται εύκολη στην εφαρμογή της, αλλά υπάρχουν πολλά θέματα. Για παράδειγμα, ο παραδεκτό, το, το παραδεκτό ημί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, θα απορρίψει ε, αιτήματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την ε, πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη, για παράδειγμα. Αυτά θα τα απορρίψει. Ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί ο, ο, ο, η σοβαρότητα, αν θέλετε, του αιτήματο ε, όσον αφορά τι υπογραφέ τώρα. Ε, εδώ πρέπει να δούμε ε, τη συγκεκριμένη κατανομή κτλ. Έχουμε διάφορες προτάσεις. Αναφέρεται το 1 εκατομμύριο πολιτών. Επίσης, ποιος, ποιος, ποιος οργανώνει τις ε, πρωτοβουλίες αυτές. Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα. Μόνο τα φυσικά πρόσωπα, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ε, καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμα, τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και πόσο χρόνο πρέπει να δίνεται ω δυνατότητα για τη συλλογή υπογραφών. Εδώ και εδώ οι απόψει δίστανται. Στη συνέχεια, όσον αφορά την υπογραφή. Ε, υπογραφές επί χάρτου. Ε, και αυτό το θέμα πρέπει να εξεταστεί. Και για οικολογικούς λόγους όμως. Όσον αφορά δηλαδή, τις υπογραφές στο χαρτί. Ε, και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ακολουθήσει μια οικολογική πολιτική και πώ θα περιορίσουμε τις υπογραφές. Για θυμηθείτε. Ε, ε, 15 χρόνια ε, ε, που είχαμε όσον αφορά την εμπειρία μας ε, και με το θέμα Λαμασούρ. Για σκεφτείτε λίγο τι ακριβώς είχε γίνει. Να δούμε λοιπόν και εδώ τι θα πρέπει να προταθεί και κατά πόσον θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε κάπως την τακτική που ακολουθούμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να πούμε ότι το καθήκον του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και να δημιουργήσει τα κατάλληλα πλαίσια. Έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η ενεργό συμμετοχή. Επίση, αποστολή μα είναι να φτάσουμε στον πολίτη. Να καταλάβει ο πολίτη ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, ε, Όσον αφορά τη δική μας τη γνωμοδότηση, πρέπει να δούμε πώς θα την διαθρώσουμε. Γιατί δεν θέλουμε απ' την άλλη να βομβαρδίσουμε την Επιτροπή με μη ρεαλιστικές ιδέες και μη επικοδομητικές ιδέες. Αντίθετα, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε την δυνατότητα αυτή έτσι ώστε να, υπάρχουν, να υπάρξουν νέες ιδέες, να υπάρξει μια νέα δυναμική, ε, να υπάρξουν κέντρα δραστήρια τα οποία να δώσουν ε, μια νέα όφηση στην Ευρωπαϊκή ε-, Ένωση. Ε, πρέπει λοιπόν εμεί να αποτελέσουμε τη γέφυρα επικοινωνία με του Ευρωπαίου πολίτε. Κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξή. Να διατηρήσουμε ζωντανό ό,τι ήδη υπάρχει. Παράδειγμα, τα κέντρα τα οποία ήδη λειτουργούν και είναι αποτελεσματικά έτσι ώστε να προωθήσουν και αυτά ε, την ε, ε, πρωτοβουλία των πολιτών, να διαδραματίσουν απόλυτα το ρόλο που του αρμόζει τα κέντρα αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν και είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, Αυτά ήθελα να σα πω σαν μια πρώτη επαφή και τώρα είμαι στη διάθεσή σα για να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Κυρία Χανίμπολ, ευχαριστώ. Η κυρία Ναλόβα δεν μπόρεσε να παραβραθεί και μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της. Θα σας πω λοιπόν αυτά που ήθελε να πει αυτή. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρμοδιότητά μας ως Επιτροπή. Και το βασικό είναι η επικοινωνία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την συζήτηση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δεν πρέπει να υπάρξουν πολλοί περιορισμοί και γραφειοκρατία γιατί θέλουμε να συμμετέχουν πολλοί πολίτες στην πρωτοβουλία να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος και όχι να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο διεθνών οργανώσεων που γνωρίζουν πώς να λειτουργούν εν μέσω γραφειοκρατίας. Εμείς θέλουμε ένα όργανο που θα μας επιτρέψει να δώσουμε φωνή στους πολίτες και τους μικρότερους οργαν... τις μικρότερες οργανώσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους διοργανωτές ε, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σημείο επαφής και επίσης θα έπρεπε να εγκριθεί ένας μηχανισμός όπου θα μπορούν όλοι να καταχωρούνται για να μπορούν να υπογράφουν. Επίσης πρέπει να υπάρξουν μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν καλύτερα την πρόταση. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρξουν μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες τις επίσημες και επίσης όταν έχουμε προτάσεις που αφορούν ε, μειονότητες ε, να μεταφράζονται και στις ε, αντίστοιχες γλώσσες. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των νέων. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε την πρόσβασή τους θέλουμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Έχουν και αυτοί το δικαίωμα να συμμετέχουν. Γι' αυτό προτείνουμε να μειωθεί η ελάχιστη ηλικία στα 16 χρόνια. Γνωρίζω ότι σε κάποια κράτη επιτρέπεται να ψηφίζουν και οι 16χρονοι. Άρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και εδώ και νομίζω ότι έτσι θα ενθαρρύνουμε περισσότερο τους νέους να συμμετέχουν και στις πρωτοβουλίες και γενικά στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να αυξήσουμε το δημοκρατικό κομμάτι στο με το να μειώσουμε τον ελάχιστο απαιτούμενο συμμετοχό των κρατών μελών στο 1 τέταρτο των μελών, δηλαδή 7 σήμερα. Και ως ε, το δημοκρατικό όργανο που λογοδοτεί στον λαό της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της πρωτοβουλίας και ότι πρέπει να ενδιαφερθούν για την πρωτοβουλία αυτή οι πολίτες. Και για να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια κριτήρια παραδεκτού, αν θέλετε. Για παράδειγμα, να έχουμε ένα ελάχιστο 5.000 υπογραφών. Αυτό πρότεινε ο εισηγητής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και συμφωνούμε με αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βερζιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ πλήρως με την εισαγωγή που έγινε και να πω ότι έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα με εσάς. Γενικά συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Ε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί ήδη οργανώσει μια συνάντηση για να συζητήσουμε το θέμα. Νομίζω ότι προκύπτει κάποια συνένεση. Βεβαίως πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Και στην πράξη θα είναι μηδενικές. Οπότε κινητοποιούμε τους πολίτες και στο τέλος τι γίνεται, ενδεχομένως να ασχοληθεί με το θέμα η Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν ένα ευέλικτο σχήμα που θα επιτρέπει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να συμμετέχουν. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα παιδαγωγικό μέσο γνωρίζουν έτσι οι πολίτες ποιες είναι οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού μπορούν να παρέμβουν. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα αφορά βεβαίως την Επιτροπή μας, γιατί η Επιτροπή μας ασχολείται με θέματα πολιτικής αγωγής, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να μειώσουμε το όριο ηλικίας γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο πολιτικής αγωγής. Και επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν πραγματικές συνέπειες, δεν νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε γραπτές υπογραφές κτλ. Έτσι θα αποφύγουμε και πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το πιο απλό μέσο που έχουμε για τις υπογραφές. Τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία να το χρησιμοποιήσουμε ως μέσο πολιτικής αγωγής, ως μέσο δημοκρατικής συμμετοχής και επικοινωνίας και θεωρώ ότι πρέπει να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα ως το μοναδικός δημοκρατικός θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την παρουσίαση και συμφωνώ και με το γεγονός ότι το πλέον κατάλληλο όργανο για την, πρωτοβουλία των, ε, της, για την ε, πρόθεση πρωτοβουλία αυτή των πολιτών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμεί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διάβλο που έχουμε στη διάθεσή μα για να προωθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει δέσμευσή μα. Ε, το οφείλουμε αυτό στον πολίτη. Και ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε ε, για να μην ε, ε, δημιουργήσουμε μέσα που στην πράξη να διαβρώνουν την δυνατότητα αυτή της πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, έχουμε και την ηλεκτρονική υπογραφή. Γιατί κοιτάξτε, πολλά είναι τα κράτη-μέλη που δεν ζητούν αυτούς τους τόνους χαρτιού. Άρα λοιπόν, γιατί να μην εξοικονομήσουμε το χαρτί όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και να μην έχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής. Επίση, όσον αφορά τη διαδικασία, η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ιδιαίτερα ε, ποιοτική. Να μην είναι ένας χώρος ε, όπου ακούγονται τα πάντα, έτσι. Πρέπει να υπάρξει μια εγγύηση για μια ελάχιστη ποιότητα. Και ένα ελάχιστο όριο ε, συλλογή υπογραφών. Παράδειγμα 40.000. Γιατί αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει Ω εγγύηση Ποιότητα αν θέλετε και νομικής ε, ασφάλειας. Θα μπορούσε λοιπόν να σκεφτεί ε, αυτό ε, η Επιτροπή, γιατί και όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια ενό πνεύματο προώθηση ω των δυνατόν περισσότερων πολιτών. Μαρκ Κλάρκιν, κοιτάξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα καλύψουμε κάπω το δημοκρατικό έλλειμμα που το οποίο υπάρχει. Έχουμε όμω κάποια προβλήματα με το χρόνο, με, με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Είναι ιδιαίτερα επαχθή στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι θα πρέπει να ελαφρύνουμε κάπω κάπω τη διαδικασία ε, και να είμαστε πιο φιλικοί προ το χρήστη. Εδώ στη τελευταία ανάλυση τι θέλουμε, να ακούσουμε του ε, ψηφοφόρου μα, ε, του ανθρώπου που εκπροσωπούμε. Άρα λοιπόν είναι πολύτιμο εργαλείο. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα φραγμό όσον αφορά το και εμπόδια, παράδειγμα, αναφορά ρυθμού ταυτότητα κτλ. Δεν πρέπει να δημιουργούμε εμπόδια και να είμαστε ιδιαίτερα διαφανεί. Και η Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα διαφανή ε, όσον αφορά την εξέταση του παραδεκτού ή μη. Αν απορρίπτει κάτι, να προβλέπεται και δυνατότητα προσφυγή. Αν δηλαδή έχουν ε, ε, συλλεγεί 300.000 υπογραφέ κτλ. Το θέμα είναι να, να ακούσουμε αυτού που συγκεντρώνουν τι υπογραφέ. Και στη τελευταία ανάλυση, τι θα γίνει στην πράξη. Αν τελικά έχουμε αυτό το 1 εκατομμύριο των υπογραφών και έχει εγκριθεί το παραδεκτό, τι θα γίνει στη συνέχεια. Πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα. Γιατί πρέπει να δώσουμε την εντύπωση πραγματικά ακούμε. Όχι δηλαδή ότι γίνονται όλα αυτά και τελικά δεν οδηγούν πουθενά. Διαφορετικά δεν θα είμαστε αποτελεσματικοί. Yeah. Τσβέρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο ε, για τον οποίο θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε με την πρωτοβουλία αυτή. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο αυτό ε, γίνεται πραγματικά δημοκρατική κοινότητα δεν ε, είναι βέβαια ανάλογη με ένα κράτο. Αλλά οι πολίτε, το θέμα είναι ότι οι πολίτε μπορούν να συμμετάσχουν στην ε, δημοκρατική διαδικασία και μέσω των εκλογών, εκλέγοντα ε, το κοινοβούλιο, τον πρόεδρο, να συμμετέχουν σε δημοψηφίσματα και να υποβάλουν νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Προτάσει για νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Η συνθήκη Λισαβόνα, λοιπόν, προβλέπει αυτό το τρίτο στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκα, τη δυνατότητα πρωτοβουλία. Όλα τα σχόλια που ακούσαμε. Ε, συμβάλλουν προ την κατεύθυνση τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη. Και ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου διανύουμε οικονομική, χρηματοπιστωτική και πολιτική κρίση. Όταν όμω ε, ε, ξεσπάει μια κρίση, τότε οι πολίτε χάνουν την εμπιστοσύνη του στους θεσμού και στους δημοκρατικού θεσμού. Ακριβώ γι' αυτό πιστεύουμε, βλέπουμε ότι δημιουργούνται αντιδημοκρατικά κινήματα, νεοναζιστικά κινήματα κτλ. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την, την υφιστάμενη κρίση και να ε, ε, ταράξουν τα θεμέλια της δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κοιτάξτε, φαίνεται ότι ζούμε ε, σε μια περίοδο υπαναχώρησης και αποστοδρόμησης και στον τομέα της δημοκρατίας και δεν οδεύουμε προς τα εμπρός. Ε, στο, υπήρξε μια έρευνα στον Economist όπου φάνηκε σαφώ ότι η υποστήριξη για τη δημοκρατία μειώνεται. Μα ακριβώ γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και εδώ υπάρχουν ορισμένα προβλήματα όμω. Η Επιτροπή προσπαθεί να περιπλέξει τη διαδικασία ώστε να τον γίνεται. Ε, δεν είναι καλό αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε αποφάσει για το παραδεκτό ή μη τη πρωτοβουλία. 300.000 πρωτοβουλίε, ε, ε, υπογραφέ κατά την άποψή μου, είναι υπερβολικό νούμερο. Δεν είναι, είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ε, θα πρέπει να έχουμε, ε, το, ε, ε, ε, να προβλέπουμε το 1 τρίτο για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία. Το 1 τρίτο των 400.000. Επίση, όσον αφορά το, το, το, το γεγονό ότι θα πρέπει να συμμετέχει το 1 τρίτο του αριθμού των κρατών μελών. Δεν είναι και καλό, αλλά δεν είναι και κακό αυτό. Γιατί Εάν ε, ε, με τέτοια κριτήρια ε, ως προς το παραδεκτό, τελικά θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που θα συμμετέχουν όλοι οι πολίτες και όχι μόνο μια ομάδα πολιτών από την ίδια περιοχή. Θέλω να ε, ε, τονίσει ιδιαίτερα η γνωμοδότηση ε, ότι πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα. Αντίθετα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο να απλοποιήσουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Νεβεντάλοβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε και ο προηγούμενο συνάδελφο, ο κύριο Βέσσερ. Ε, 300.000 είναι πάρα πολλέ. Ή 50.000 ή 100.000 αρκούν. Όμως ε, προκύπτει το εξή ερώτημα. Ε, το πρώτο ε, κατόφλι θα είναι 50.000. Ε, τώρα να φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα θα πρέπει να ε, υπάρξει ένα όριο. Και, αλλά αυτό, εδώ πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το πρωτογενέ δίκαιο. Παράδειγμα, αλλαγή τη έδρα ε, στο Στρασβούργο. Ε, κατάργηση του Στρασβούργου. Ε, αυτό είναι θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη. Και εδώ πρέπει να το δούμε. Και να δούμε όμως τι δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην πρωτοβουλία των πολιτών. Με άλλα λόγια, να δούμε τι θα συμβεί. Ας πούμε δηλαδή ότι συγκεντρώνεται ο επαρκής αριθμός πληροφοριών. Να δούμε το επόμενο βήμα. Θα έχουμε κανονισμό ή κάτι άλλο. Πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό. Elnök asszony, tisztelt kollégák, csak egyet érteni tudok. Συνάδελφοι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον κύριο Ζελ που ζήτησε να αυξηθεί η δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αυξηθεί ο ρόλος, το βάρος, το ειδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί οι ευρωβουλευτές είναι το καλύτερο σύμβολο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Πρόσφατα εγκρίθηκε ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την εξορρυκτική βιομηχανία και τη χρήση κιανίου. μετά την περίεργη ψηφοφορία η Επιτροπή αναθεώρησε την πρότασή της και η νέα πρόταση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Πρόταση η οποία ναι, έλεγε ότι μπορεί να συνεχιστεί η εξόριξη με χρήση και ανίου Αυτό δεν είναι παρά ένα παράδειγμα. Δείχνει ότι το Κοινοβούλιο αποτελεί το μοναδικό σύμβολο και αν τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα είναι αυτά που υπαγορεύουν τις αποφάσεις αντίθετα στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για δημοκρατικό έλλειμμα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο είναι το καλύτερο μέρος όπου θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος της πρωτοβουλίας των πολιτών. Λοιπόν, Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την κυρία Ρόζα Τούν να εργαστεί με την ησυχία της. Εγώ προσωπικά έχω να σας πω ότι έχω σημαντικές επιφύλαξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, όσον αφορά τις απογοητεύσεις που θα δημιουργήσουμε με κάτι τέτοιο. Όλοι όσοι θα συμμετάσχουν θεωρούν ότι στο τέλος θα υπάρχει ένας νόμος και θα διακανονιστούν τα πράγματα όπως θέλουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στη δημοκρατία. Αυτό είναι το πρόβλημα εγώ έχω ένα πρόβλημα με το θέμα. Όχι επειδή είμαι κατά τη συμμετοχή των πολιτών, αλλά επειδή ξέρω ότι ε, θα δημιουργήσουμε πολλέ προσδοκίε. Έχω έναν συνάδελφο που μαζεύει υπογραφέ, δεν ξέρω, για να μην εργαζόμαστε την Κυριακή, κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρω ότι κάτι που έχουμε στο Κοινοβούλιο συνεχώς αυτές τις ε, γραπτές δηλώσεις που υπάρχει στο Κοινοβούλιο. Εγώ δεν υπογράφω καμία από αυτές γιατί θεωρώ ότι η εργασία μου είναι να εργάζομαι εδώ στο σώμα, να προετοιμάζω την νομοθεσία μέσω των ε, ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών και όλη αυτή η πλημμύρα των γραπτών δηλώσεων έρχεται και μου λέει υπογράψε εδώ, υπογράψε εκεί, δεν υπογράφω τίποτα ακόμα και αν συμφωνώ με την ιδέα γιατί θεωρώ ότι έτσι δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Λοιπόν, ελπίζω η κυρία Τούν να καταφέρει να συμβάσει τα πράγματα, να έχει στο τέλος κάτι βατό που δεν θα μας δυσκολεύσει τη ζωή περισσότερο από είναι ήδη δύσκολη σήμερα. Πολύ επιλεκτική. Αν θέλετε να πεις κάτι ρόζα, πάντως παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Και εγώ έτσι τα βλέπω τα πράγματα, δυστυχώς. Ε, με συγχωρείτε, θα μιλήσω καλύτερα ε, πολωνικά. Γιατί, όπως σας είπα, συμφωνώ με εσάς και για να μην περιπλέξω τα πράγματα περισσότερο, έχω να σας πω ότι διάφορα θέματα δεν τα έχω θίξει καν που υπάρχουν εκεί. Προστασία δεδομένων, τι θες κάνουμε αυτές τις υπογραφές, θα τις διατηρήσουμε κάπου ή όχι. Πόσες πληροφορίες θα αναφέρονται Υπάρχουν διαφορετικά έγγραφα. Η Κομισιόν θα τα απαριθμίσει. Τι θα γίνει με εκείνους που ζουν εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες. Γιατί τα εκλογικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παραδείγματο χάρη σε ορισμένε χώρε ψηφίζουν οι 16χρονοι, σε άλλοι μόνο οι 18χρονοι. Τι γίνεται με εκείνου που έχουν δικαίωμα ψήφου σε μια χώρα, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε μια άλλη χώρα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, είμαι σίγουρη. Και θεωρώ όμως ότι εάν υπάρχει καλή βούληση θα μπορέσουμε κάτι να καταφέρουμε. Και παρόλο στις δυσκολίες θα έπρεπε νομίζω η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών να θεωρηθεί σαν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία η οποία θα δώσει στους πολίτες δυνατότητα να κατανοήσουν ότι είναι πολίτες με δυνατότητα παρέμβασης στην νομοθεσία. Είναι μια πρόκληση για όλους εμάς εδώ και για το Συμβούλιο βέβαια. Γιατί το Συμβούλιο προετοίμασε ένα διαφανές έγγραφο, αλλά στρεφόμαστε και προς την Κομισιόν. Χρειαζόμαστε στενή συνεργασία. Πρώτος, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση του θέματος αυτού. Καλή διασκέδαση σου εύχομαι και αποτελεσματικό στην προετοιμασία ενό λογικού εγγράφου. Περάμε στο σημείο 11 τη μιλήσια διάταξη. Έγκριση των ε, αποφάσεων τη Κομισιόν. Το πήρατε απόψε. Συμφωνήσατε, φαντάζομαι. 12 στα διάφορα. Κάποιο άλλο νομίζει ότι κάτι πρέπει να πει. Όχι. Ωραία. Σα εύχομαι λοιπόν καλέ διακοπέ. Εύχομαι και ο διερμηνεί. Και θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Γεια σας.